Καλημέρα. Ξεκινάει η συνεδρίαση. Ξεκινάμε με το σημείο 7 της ημερήσιας διάταξης. Ε, πρόκειται για την ανάλυση που έχει κάνει η Διφιντεύκο. Ε, υπάρχει μια επιστολή από τους επίτροπους Χάρκε Μίμητσε, από... δυστυχώς ε, δεν δεν το είπαν όλοι. Δεν το είδαν όλοι. Δικό μου είναι το λάθος. Ζητώ συγγνώμη. Αλλά βέβαια και εγώ εχθές το πήρα το έγγραφο και δεν μπόρεσα να το δώσω και σε κανέναν άλλον. Να σας χαιρετήσω λοιπόν. Ε, και τις δύο γενικές διευθύνσεις να σας ε, δώσω και τη δυνατότητα να παρουσιάσετε το έγγραφο. Ποιος ξεκινά, η Τεύκο παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, θα μιλήσω γαλλικά. Σας ευχαριστώ που διοργανώσατε αυτή τη συνάντηση. Είχαμε ήδη τη δυνατότητα να μιλήσουμε για τα αποθέματα που ε, είχε στη διαχείρισή της η ΔΕΦΚΟ το 2016. Όπως είπατε, μίλησαμε και με τον Επίτροπο Μίμητσα μέσα στην διαδικασία απαλλαγής για το 2016. Αυτή η συνάντηση παρόλα αυτά είναι χρήσιμη, γιατί θέλουμε να μιλήσουμε για την επίδοση στο θέμα της ε, οικονομικής διαχείρισης. Καταρχάς να θυμίσω ότι αυτά που μιλάμε, αυτά που λέμε EAMR, δηλαδή External Assistant Management Report στα αγγλικά, στην ουσία ε, είναι εκεί για να ε, υποστηρίξουν τη δήλωση εξοπιστίας των επικεφαλής ε, των αντιπροσωπιών σύμφωνα με το άρθρο 67,3 του Δημοσιονομικού Κανονισμού ο οποίος ζητά από τους επικεφαλής των αντιπροσωπιών με μια τέτοια δήλωση να υποδείξουν ότι έγινε με νόμιμο και σωστό τρόπο η διαχείριση των κονδυλίων και σύμφωνα με τους στόχους της εφαρμογής της ε, συνεργασίας για την ανάπτυξη. Πάμε όμως λίγο πιο πέρα από αυτή την απλή δήλωση. Θέλαμε να φτιάξουμε ένα πραγματικό εργαλείο ελέγχου της διαχείρισης των κονδυλίων που θα μας επιτρέψει ένα monitoring σε πραγματικό χρόνο γιατί υπάρχει ένα σύστημα πληροφορικής και είναι και το θαύμα της πληροφορικής σήμερα που μας επιτρέπει να βλέπουμε μέρα με τη μέρα ε, την εξέλιξη των KPIs. Χρησιμοποιούμε λοιπόν αυτό το σύστημα σε κεντρικό επίπεδο αλλά και σε όλα τα στάδια και τα εισβαθμίδες της οργάνωσης. Τα EAMR πέρα από αυτούς τους KPIs, τους δείκτες ε, δηλαδή επιδόσεων, καλύπτουν και κάποια άλλα στοιχεία, τα οποία μας επιτρέπουν να έχουμε μια αξιολόγηση της διαχείρισης ε, της ε, συνεργασίας. Τα σημεία που καλύπτονται είναι ο πολιτικός διάλογος, η εταίροι τα αποτελέσματα ε, που έχουν επιτευχθεί σε επίπεδο συνεργασίας, οι κίνδυνοι που ε, εντοπίζονται από την αντιπροσωπεία και ποια είναι τα μέτρα που έχουν ληφθεί για τον περιορισμό των κινδύνων, ποια είναι τα μέτρα που βελτιώνουν την ορατότητα των προγραμμάτων, πώς ε, ε, χρησιμοποιείται και η, ε, πώς ε, διασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα της, των επιχορηγήσεων γενικά και όλα τα στοιχεία των επιχορηγήσεων, γενικά ε, μία αξιολόγηση του συστήματος εσωτερικού ελέγχου και της αποτελεσματικότητας των ιστορικών ελέγχων και των εξωτερικών ελέγχων των συστημάτων. Επίσης, ε, ε, υπάρχουν σχόλια σχετικά με τη διαχείριση των ανθρωπίνων πόρων και στο τέλος μια σύνοψη των KPIs και μία δήλωση αξιοπιστίας του επικεφαλής της αντιπροσωπείας. Έτσι λοιπόν, ε, προσπαθούμε να δώσουμε κάποιες οδηγίες σχετικά με τη σύνταξη των εκθέσεων αυτών των EAMR. E ε, αυτό γίνεται το Δεκέμβρη, το Γενάρη υπάρχει υπογραφή των εκθέσεων, το Φλεβάρι οι διευθυντές ε, συντάσσουν μία έκθεση ε, βάσει αυτών των εκθέσεων των επικεφαλής των αντιπροσωπιών, οι διευθυντές, και το Μάρτι ε, υπογράφεται η δήλωση αξιοπιστίας και γίνεται και μια έκθεση για το Κολέγιο των Επιτρόπων. Τον Μάιο διαβιβάζουμε το σύνολο των πληροφοριών στα άλλα θεσμικά όργανα, ε, Κοινοβούλιο, Συμβούλιο, ελεγκτικό συνέδριο. Τον Ιούνιο του 2017 το Κολέγιο των Επιτρόπων ενέκρινε την ετήσια έκθεση της Επιτροπής και το σύνολο των πληροφοριών, των αναλυτικών πληροφοριών δίνεται στο Κοινοβούλιο είτε το Μάιο με ένα αρχείο Excel ή τον Οκτώβρη ή Νοέμβρη ως ανάλυση των αποτελεσμάτων του έτους 2017. Όπως ε, έλεγα, είναι δύο οι στόχοι για αυτή, σε αυτή την έκθεση των επικεφαλής των αντιπροσωπιών. Καταρχάς, η δήλωση αξιοπιστίας. Είναι πολύ σημαντικό η έκθεση στην ουσία της να έχει ε, όλα τα στοιχεία που επιτρέπουν στους επικεφαλείς να υπογράφουν με τα λόγου γνώσεως ε, και οι πληροφορίες που υπάρχουν σε αυτή την έκθεση θα πρέπει να είναι πραγματικές και αξιόπιστες. Το σύνολο των μέσων που είναι διαθέσιμα, δηλαδή οι δημοσιονομικοί πόροι και οι ανθρώπινοι πόροι, θα πρέπει να φαίνεται ότι χρησιμοποιήθηκαν για τους ε, δεδηλωμένους στόχους, σύμφωνα με την αρχή της καλής ε, δημοσιονομικής διαχείρισης και η δήλωση καταλήγει λέγοντας ότι οι εσωτερικές διαδικασίες ελέγχου της αντιπροσωπείας εγγυώνται την νομιμότητα και την ε, σωστή, τη χρηστή διαχείριση των ε, συναλλαγών. Επίσης, ως προς τον ε, έλεγχο διαχείρισης των KPIs, έχουμε έναν ε, έλεγχο πραγματικού χρόνου αυτών των δικτών σε όλα τα επίπεδα, σε επίπεδο αντιπροσωπείας, διεύθυνση και γενικής διεύθυνση. Διασφαλίζουμε ότι πέρα από αυτό το μόνιμο monitoring έχουμε μία έκθεση τουλάχιστον κάθε τρίμηνο η οποία θα μπορεί να συζητείται στην Διοικητική Επιτροπή της ΔΕΦΚΟ και βάσει αυτού λαμβάνουμε μέτρα ε, ως προς τις αντιπροσωπείες ή τους ειδικού δείκτες, δηλαδή μέχρι το τέλος του έτου θα πρέπει η κατάσταση να μπει ε, στη σωστή ροή αν υπάρχουν σημαντικές αποκλήσεις. Ως προς τη διαφάνεια, οι δείκτες ε, υπάρχουν στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων, τον απολογισμό δηλαδή της DigiDefco και DigiNear, εδώ να παρεκκλίνω λίγο και να πω ότι μετά από τις ε, συζητήσεις με τον Επίτροπο Μίμητσα κατά τη διαδικασία της απαλλαγής ξανά εξετάσαμε τις ε, συνθήκες ε, μετάδοση αυτών των πληροφοριών και δεδομένων στο Κοινοβούλιο. Μάλλον ήταν πολύ περιορισμένη και στενή η ερμηνεία της εμπιστευτικότητας. Έτσι λοιπόν σε αυτό το φάκελο δεν αποκαλύπτουμε στοιχεία τα οποία μπορεί να βλάψουν τις ε, σχέσεις μας με τις τρίτες χώρες. Βέβαια, ε, το 99% των πληροφοριών σε αυτές τις εκθέσεις είναι ε, δημόσιες πληροφορίες. Οπότε καλό θα είναι να γίνει μια, ένα ξεκαθάρισμα, να με, δημοσιοποιηθούν οι εκθέσεις για το 2017 και χωρίς τα προβλήματα της εμπιστευτικότητας ε, να δίνονται στο Κοινοβούλιο για να τις χρησιμοποιείτε χωρίς κανένα περιορισμό. Χωρίς αμφιβολία είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε αναλυτική ανάλυση. Τα συνολικά αποτελέσματα για το 2017 ανά αντιπροσωπεία δείχνουν ότι τα αποτελέσματα είναι καλά. Δηλαδή στις 108 αντιπροσωπείες που πρέπει να συντάξουν έκθεση, 101 επιτυγχάνουν τα αποτελέσματα, αποτελέσματα που ε, ανέρχονται σε πάνω από το 60% των KPIs. Δηλαδή μόνο 7 είναι οι αντιπροσωπείες που δεν μπόρεσαν το 2017 να επιτύχουν το 60% των KPIs. Και τώρα δίνω το λόγο μου στον συνάδελφο Μακ Τζόνστον για τα αναλυτικά αποτελέσματα σχετικά με τη Γενική Διεύθυνση NEAR. Ευχαριστώ όλους, σας ευχαριστώ πρόεδρε, να ευχαριστώ και για την ευκαιρία που μας δίνετε να παρουσιάσουμε τα αποτελέσματα για το 2016 από τη δικιά μας Γενική Διεύθυνση. Πρόκειται για τη δεύτερη περίπτωση στην οποία η DGN αναφορά, δίνει αναφορά για τα ΚΠΑ στην πρώτη φορά ήταν για το 2015. Αυτό αποτέλεσε λοιπόν και εντομία και φυσικά η, η Γενική μας Διεύθυνση δημιουργήθηκε αρχές 2015 από, γενική, από διεύθυνση της ΔΕΦΚΟ και από την παλιά Γενική Διεύθυνση Διεύρυνσης. Και έτσι λοιπόν Αναφέρουμε για 18 KPIs και φυσικά γνωρίζουμε και γνωρίζαμε ότι το Κοινοβούλιο ήθελε να σχολιάσουμε και να κάνουμε αναφορά και για 24 KPI. Αυτό και κάναμε και το 2016. Να σας πω ότι μάθαμε στον δρόμο λίγο. Πρόκειται για μια διαδικασία να εξελίξει. Θεωρούμε ότι προχωράμε γενικά χρόνο με το χρόνο και ελπίζουμε ότι τα πράγματα θα βελτιωθούν και το 2017 του χρόνου. Να δούμε τι έχουμε πετύχει λοιπόν, συνολικά. Νομίζουμε ότι τα αποτελέσματα είναι αρκετά θετικά τα απορίσματα. Θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι υπήρξε και κάποια βελτίωση για το ότι 20 από τα KPIs λοιπόν, από τα 24 στο σύνολό τους, αν κοιτάξουμε τα ενοποιημένα αποτελέσματα του 2016, πετύχαμε το στόχο σε επίπεδο γενική διεύθυνση. Αυτό σημαίνει επίπεδο επιτυχίας 83% η απόδοση το 2016 είναι συγκρίσιμη με το 2015 όπου και αναφέραμε για 18 KPIs και πετύχαμε τα, τους στόχους μας, τα benchmarks για 12 από αυτά, 87%. Ας κοιτάξουμε τώρα ποιες αντιπροσωπείες δεν πέτυχαν τα benchmarks το 60% για τα KPIs και πάλι βλέπουμε ότι οι τάσεις είναι ενθαρρυντικέ. Αυξάνονται οι προσωπίες που πετυχαίνουν τους στόχους για τα πιο πολλά KPIs το 2016. Στα τέλη του 2016 προσμετρήσαμε λοιπόν για 22 αντιπροσωπείες στα KPI και μόνο μία εξ αυτών δεν είχε πετύχει τον στόχο του 60% των KPI και αυτή η αντιπροσωπεία είναι η Συρία. Αυτό δεν προκαλεί φυσικά εντύπωση. <clears throat> Κοιτώντας λοιπόν τώρα τις διάφορες κατηγορίες KPI, βλέπουμε ότι στις τρεις κατηγορίες έχουν σημειωθεί βελτίωσεις. Κοιτώντα λοιπόν την ε, καλή χρηματοοικονομική διαχείριση και την αποτελεσματική χρήση των πόρων για το KPI 1, βλέπουμε βελτίωση. Άρα η αρχική πρόβλεψη πληρωμών ήμασταν 99% ακριβείς το 2015 ή το 2016 δε το ποσοστό εγκυρότητας ήταν 97%, 95% και το KPI υπαριθμών 7 μειώθηκε κατά 33% 679 εκατομμύρια από 2 δισεκατομμύρια τον Ιανουάριο σε 1,4 δισεκατομμύρια το Δεκέμβριο του 2016. Παρομοίως ε, το παλιό ραλ KPI ε, 9 περιορίστηκε κατά 376, 376 εκατομμύρια. Στη συνέχεια, να δούμε τα Project Traffic Lights. Αυτά τα δύο KPIs δεν τα συμπεριλάβαμε στην αναφορά του 2015, ήταν καινούριο το στοιχείο αυτό του 2016. Κοιτώντα λοιπόν το υπαριθμό 5 και 6, βλέπουμε ότι προφανώς είναι μέλλοντος τράφι και προφανώς ε, χρειάζεται πλήρης ε, χρήση των πόρων για να πετύχουμε τα αποτελέσματα στα τέλη του έργου. Κοίτατο λοιπόν τι έχουμε πετύχει. Διαπιστώνουμε το ότι το σύνολο των έργων το οποίο χαρακτηρίζεται ως προβληματικό είναι 36% της συνολικής αξίας των έργων και από 2.149 έργα, 576 ήταν εκείνα, 27% τα οποία θεωρούνται προβληματικά, τα οποία χαρακτηρίζονται προβληματικά. Μία μικρή παρένθεση στο σημείο αυτό, γιατί φυσικά το benchmark έχει να κάνει με έργα που έχουν κόκκινο φως, έχουν λάβει κόκκινο φανάρι, όχι προβληματικά απλά. Τα προβληματικά είναι, αν θέλετε, αυτά τα οποία είναι κόκκινα και πορτοκαλί. Κοιτώντα ε, τα benchmarks, ε, ε, είμαστε εντό των ορίων και για το KPI 5 και για το KPI 6. Θα έλεγα ότι έχει γίνει σχετική ανάλυση και αυτό που διαπιστώσαμε είναι ότι σε διάφορες περιπτώσεις, όταν κοιτώντας προβληματικά τέτοια έργα, εικάζουμε ότι η αρχική πρόβλεψη ήταν υπερβολικά αισιόδοξη. Άρα θα πρέπει να μπει μια νότα ρεαλισμού σε σχέση με το τι μπορεί πραγματικά να πετύχει το κάθε έργο. Και θα ήθελα φυσικά να αναφέρω ότι λειτουργούμε σε κάποια τμήματα του κόσμου όπου οι συνθήκες είναι ιδιαίτερω δύσκολες. Όταν λοιπόν αντιμετωπίσαμε τις δυσκολίες αυτές, όταν αντιμετωπίζουμε δυσκολίε, προβαίνουμε διορθωτικά μέτρα, αλλάζουμε και το σχεδιασμό των έργων, αν είναι απαραίτητο. Δεν θα ξέρουμε λοιπόν μέχρι τα τέλη του χρόνου, μέχρι την αναφορά στα τέλη του χρόνου το πώς εξελίσσεται η κατάσταση και ποια είναι η τάση σε ό,τι αφορά τα προβληματικά αυτά έργα, σε ό,τι αφορά την ετήσια δραστηριότητα για το 2017. Εξετάζοντα τώρα το επόμενο, την επόμενη ομάδα και το KPI, την αποτελεσματικότητα των ελέγχων συγκεκριμένα, διαπιστώνουμε ότι είναι αυξημένη η αποδοτικότητα των ελέγχων και εδώ και εξετάζοντας τα KPI οι 12 έως και 20 διαπιστώνουμε ότι για παράδειγμα το 2016 ο αριθμός των πληρωμών των χρηστήτως των πληρωμών που αποτράπηκε από ελέγχους εξάντα ήταν 4,64%. Και έτσι λοιπόν εντοπίσαμε μεγαλύτερο ποσοστό των προβλημάτων σε επίπεδο εξαντέκ των προτέρων ε, σε σχέση με το προηγούμενο έτος και παρομοίως κοιτώντα ε, τα τελευταία ομάδα KPI ε, ό,τι αφορά την εκτέλεση των ετησιων ελεγχών 29 και 24. Διαπιστώνουμε ότι έχουμε τρία πράσινα KPI το 2016, ενώ το 2015 το αντίστοιχο αριθμητικό στοιχείο ήταν ένα. Ένα μόνο τέτοιο KPI πράσινο. Τώρα, να στραφούμε σε ένα πολύ σημαντικό θέμα του τι κάνουμε με όλες αυτές τις πληροφορίες σε ό,τι αφορά τα KPI, τι σκοπό εξυπηρετούν και ποια είναι η τοποθέτηση, αν θέλετε, στην Γενική Διεύθυνση στις αντιπροσωπείες. Επειδή ο έτη, λοιπόν, ασχολούμαστε με αυτή την εργασία από 18-21 KPIs και να σας πω ότι τα λαμβάνουμε πάρα πολύ σοβαρά τα KPIs στη γενική μας διεύθυνση, στη γενική διεύθυνση NEAR. Είναι μια διαδικασία λοιπόν, όπως σας είπα, να εξελίξει. Θέλουμε να εξασφαλίσουμε ότι θα γίνουν σωστά κατανοητά τα στοιχεία αυτά. Και ε, μηνιαίως ε, κάνουμε εκθέσεις για τα, για τα οικονομικά στοιχεία και εδώ αποτυπώνονται όλες οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στα dashboards. Αυτή η τύση λοιπόν άσκηση η μηνιαία οι μηνιαίες εκθέσεις ε, συζητιέται σε τακτικό επίπεδο στις, ε, στα, στην Διαχειριστική Επιτροπή. Όταν λαμβάνουμε λοιπόν τις εκθέσεις αυτές, όταν λάβαμε μάλλον την εκθέση αυτή τον Φεβρουάριο, τι κάναμε. Έγινε μια διεκπαιρετική, αναλυτική ανάλυση. Συζητήσαμε και με τους γενικούς διευθυντές, τους εκάστοτε υπεύθυνου για την γεωγραφική περιοχή και συμφωνήσαμε για τις δράσεις που έπρεπε να ληφθούν, για, τα, για τους πόρους και τα μέσα τα οποία χρειάζονται οι αντιπροσωπείες και πού θα πρέπει να εστιάσουν την προσοχή τους. Γίνονται τακτικές ε, συζητήσεις ε, για τα KPIs και τα αποτελέσματα με τους ε, επικεφαλής των λειτουργικών ομάδων στις Βρυξέλλες. Γίνονται επίσης συζητήσεις με τον επικεφαλής των αντιπροσωπιών στις αντιπροσωπείες και με τους επικεφαλείς των ε, λειτουργικών δράσεων στις αντιπροσωπείες. Την προηγούμενη, τον προηγούμενο μήνα έγινε μια τέτοια συζήτηση και ε, συζητήθηκαν και συνολικά όλες ε, οι οικονομικές συμβάσεις για την δημοκρατία της Μακεδονίας και εξετάσαμε τι θα πρέπει να γίνει από τώρα μέχρι τα τέλη του χρόνου για να πετύχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Αναφέρθηκα στο γεγονός ότι συζητούνται αυτά και σε επίπεδο υψηλότερων αξιωματούχων και τα αποτελέσματα λοιπόν ε, είναι ότι χρειάζεται τακτική επικοινωνία και από επιστολές τα οποίες αποστάλλονται στις αντιπροσωπείες και επικεντρωνόμαστε για παράδειγμα σε θέματα πλήρους εκτέλεσης ε, του αναθεωρημένου σχεδίου εφαρμογής πριν τα τέλη του έτους. Εδώ λοιπόν είμαστε σε έντονη επαφή με τι αντιπροσωπείες. Αυτά συνοπτικά σε ό,τι αφορά την γενική μα διεύθυνση, τη γενική διεύθυνση ΝΙΑ, σε ό,τι αφορά τα αποτελέσματα των KPI. ευχαριστώ. Ε, ε, ευχαριστώ. Να, μια σύνοψη της κατάστασης για τους δείκτες KPI όσον αφορά την ΔΕΦΚΟ. Και από τότε που θεσπίστηκαν αυτοί οι δείκτες βλέπουμε ότι είναι συνεχής η βελτίωση. Μα αυτό είναι φυσικό. Γιατί με τους δείκτες μπορούμε να εστιαστούμε σε συγκεκριμένα προβλήματα για τις αντιπροσωπείες. Παράδειγμα, χτυπητό είναι οι προθεσμίες ε, πληρωμών, γιατί είπαμε ότι εκεί υπήρχε ε, πρόβλημα για διαφορετικούς ε, λόγους το 16. Οπότε τώρα έχουμε ακόμα πιο δύσκολους στόχους για τις πληρωμές και με τους δείκτες KPI τώρα μπορούμε να δούμε κατά πόσον τηρούνται αυτές οι προθεσμίες για τις συμβάσεις, ε, τι γίνεται με τα τιμολόγια, εάν ε, καταχωρούνται μέσα σε μια εβδομάδα και έτσι η ΔΕΦΚΟ μπορεί να φτάσει τους μέσους όρους της Κομισιόν. Επομένως, αποδίδουν τα KPI γιατί έτσι μπορούν να στιάσουν την προσοχή τους διάφορες υπηρεσίες ε, όσον αφορά συγκεκριμένα προβλήματα που επισημαίνονται επομένως. Όσον αφορά τις τρεις κατηγορίες KPIs έχουμε διάφορες βελτιώσεις, να σε φέρω δύο, όσον αφορά την αξιοποίηση των πόρων της Ένωσης, πρώτα πρώτα την ε, μείωση των προχρηματοδοτήσεων και πήγαμε σχεδόν στο μισό και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό αφορά μία τετραετία. Και αυτό γίνεται διότι είμαστε σε ένα διαρκή αγώνα. Δηλαδή αδειάζουμε την πανιέρα αλλά γεμίζει ακόμη πιο ε, γρήγορα και αυτό το κάνουμε προσπαθώντας να μην έχουμε τη σόρευση των προγραμματοδίσεων όπως το παρελθόν. Επίσης έχουμε μείωση των παλαιών συμβάσεων όσον αφορά κάποιες ε, συμβάσεις χαρτοφυλακίου γιατί πρόκειται για δραστηριότητες που έχουν ολοκληρωθεί και εδώ από το 19 πήγαμε σε τριχόνια στο 15% και έχουμε κάποια σημαντικά μέτρα φέτος ούτως ώστε να μειώσουμε αυτόν τον αριθμό των ε, ε, συμβάσεων που έχουν ε, λήξει. Τώρα όσον αφορά τον ιστορικό έλεγχο επίσης μετρούμε τον αποτελεσματικότητα των εκτονιστέρων ελέγχων οπότε και έτσι το 17 μπορούσαμε να ανακτήσουμε 132 εκατομμύρια και αυτά τα 132 τώρα να καταβληθούν στους επιλέξιμους δηλαδή είναι 46% των ετήσιων πληρωμών είχαμε benchmark 2% και 14% ε, μη σε πληρωμές σε επιλέξιμους. Άρα, να το 2%. Άρα βλέπουμε ότι είναι σημαντική η βελτίωση όσον αφορά τα, τα προγράμματα οικονομικών ελέγχων και τώρα έχουμε ε, αυτά τα, ε, αυτούς τους δείκτες επιδόσεων που χρησιμοποιούνται. Τώρα όσον αφορά τα αποτελέσματα για τις αντιπροσωπείες Ξεκίνησαμε με 22 ε, που δεν πληρούν τους ε, στόχους ε, για το 60% των δικτών επιδόσεων που τους αναλογούν. Αυτό είναι πάρα πολύ αξιόλογο γιατί εποπτεύουμε το τι γίνεται, έχουμε συγκεκριμένα προγραμματά δράσεων, αυτά τα οποία έχει ορίσει αρμόδια γεωγραφική διεύθυνση που αναλογεί, που αντιστοιχεί τέλος πάντων γεωγραφικά στις ε, αντιπροσωπείες αυτές. Η διαχείριση δυσκόλεψε βέβαια για λόγους ασφαλείας και πολιτικούς λόγους. Και έτσι αυτοί οι δείκτες ε, ως από το πλήστον είναι στο κόκκινο. Όμως ε, αναζητούμε τις αιτίε και προβαίνουμε σε δύο Το, Όσον αφορά τώρα τα φανάρια με τα τρία χρώματα. Το πράσινο σημαίνει ότι πάνε καλά, το κίτρινο έτσι και έτσι και κόκκινο σημαίνει ότι τα πράγματα έχουν κάπως κολλήσει και Πρόκειται επομένως για ένα εργαλείο πάρα πολύ σημαντικό και το Βούλιο μας προέτρεψε να αναβαθμίσουμε την ανάλυση μας σε αυτό το μέτωπο και για πρώτη φορά το 2016 μπορέσαμε να έχουμε μια τυπολογία ε, και όσον αφορά τις καθυστερήσεις και επίσης όσον αφορά κάποια προγράμματα και έργα που δεν μπόρεσαν να καλύψουν τους τεθέντες στόχους. Επίσης, είπαμε ότι θα πρέπει να δούμε τι διορθωτικά μέτρα θα πρέπει να ληφθούν ούτως ώστε να διορθωθούν τα προβλήματα. Πολύ χρήσιμο αυτό Το θέμα της τυπολογίας γιατί έτσι εντοπίσαμε όπως είπε και ο Μάρκ ποια πρέπει να είναι η λογική της παρέμβασης και εκεί ήταν η αδυναμία των ε, προγραμμάτων των έργων κάποια μέτρα που έχουν ληφθεί για τον εντοπισμό ε, έγινε ανάλυση των ε, κινδύνων και έτσι έχουμε αντιμετώπιση πιο ρεαλιστική σε σχέση με τους ε, στόχους που πρέπει να πετύχουμε γιατί πρόκειται για κάποια προγράμματα για τα οποία υπάρχει κάποια εξασφάλιση επίτευξης τελικός των τεθέντων στόχων. Πρόκειται για 300 έργα αυτά μέσα σε δύσκολες πολιτικές συγκυρίες και θέματα ασφαλείας, δυσκολίες διαχείρισης από τους εταίρους μας, αλλά με την τυπολογία αυτή μπορέσαμε να συνδυάσουμε τις ευμέρους δράσεις. Ο στόχος ήταν να μειώσουμε τα έργα που βρίσκονται στο κόκκινο. Μιλούμε για 4%, 10% το σχετικό benchmark. Και επίσης ε, έχουμε αυτά τα οποία αφορούν και την Ευρώπη. Τέλος, όπως σας έλεγα και στην αρχή, έχουμε τους δείκτες αλλά και τα EAMR πολύ χρήσιμα και τα MEN και τα δείκτες Θα συνεχίσουμε επομένω να επενδύουμε σε αυτό το σύστημα και εδώ και ένα χρόνο, ενάμιση έχουμε αυτό το dashboard ούτως ώστε με αυτή την εργαλειοθήκη, ας την πούμε, μπορούμε να παρακολουθήσουμε ε, σαν κονσόλα, ας πούμε. Μπορούμε να παρακολουθήσουμε τι γίνεται, τι γίνεται με αυτά τα προγράμματα και να δούμε τα της διαχείρισης σε σχέση με τους στόχους. Στη συνέχεια ε, θεωρήσουμε ότι τώρα πια είναι μέσα στην κουλτούρα της ΔΕΦΚΟ οι δείκτες επιδόσεων και δεν υπάρχει και σε κάθε, σε κάθε συνάντησή μας αναλύουμε τα KPI. Και βέβαια εξελίσσεται αυτή η υπόθεση μέσα στον χρόνο γιατί ε, έχουμε τους δείκτες για να βρίσκουμε τα προβλήματα και να τα λύνουμε. Είναι κάπως σαν τα φανάρια της τροχέας. Και με αυτά ζητούμε από τους συναδέλφους πέραν ε, των στόχων ε, κάπως ε, απεσιόδοξα εξετάζουμε τι μέτρα πρέπει να ληφθούν να επισημαίνουμε ποια είναι τα προγράμματα, ποια είναι τα έργα όπου υπάρχουν κάποιοι κίνδυνοι και να μην αδιαφορούμε για αυτούς. Άρα ξέρουμε ποια στοιχεία θα μετέλθουμε για τους στόχους που μπορεί να είναι φιλόδοξοι. Σας ευχαριστώ και σήμερα είναι ιδιαίτερη ημέρα και χάρηκα ιδιαίτερος και πιστεύω ότι είναι και πάρα πολύ δίκαιο το γεγονός ότι αναφέρεται ότι πρόκειται για ένα χρήσιμο εργαλείο. Να σας ευχαριστήσω για όλη τη δουλειά που κάνετε με τα δεδομένα, γιατί εμείς ζητήσαμε την ε, δουλειά αυτή και χαίρομαι που αναφέρετε ότι είστε ευγνώμονε σε ό,τι αφορά το θέμα αυτό. Σας ευχαριστώ. Και νομίζω ότι είναι κοινό ο στόχος. Αποτελεσματικότητα και βελτίωση της αποτελεσματικότητας και σε ό,τι αφορά και τις δομές ε, διαχείρισης ε, σε ό,τι αφορά την ε, τον έλεγχο και την παρακολούθηση από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Χαιρόμαστε λοιπόν για το γεγονό ότι η DG DEFCO τα παίρνει αυτά στα σοβαρά και η DG ε, NIR έχει ξεκινήσει τη δουλειά και ελπίζω να προχωρήσει και η DG NIR να βρεθεί εκεί που βρίσκεται ήδη η DG DEFCO γιατί έτσι μπορούμε να δώσουμε λοιπόν στον κόσμο μια εικόνα του πώς ε, χρησιμοποιούμε αποτελεσματικά τα μέσα αυτά. Έχω και κάποιες ερωτήσεις να κάνω, δεν θα προκαλέσει έκπληξη. Θα ήθελα και η DG Near, όπως είπατε, να ασχοληθεί να, μεθοδικά και να προσεγγίσει τη DG DEFCO. Και η DG DEFCO μας δίνει πάντα μια ενοποιημένη, ένα, ένα ενοποιημένο κατάλογο των έργων. Ε, θα ήθελα να το κάνει αυτό και η DG NIR και αν θα μπορούσε να απλοποιηθεί και η πρόσβαση στα έργα, αυτό θα ήταν πάρα πολύ χρήσιμο. Να ξεκινήσουμε με την Γενική Διεύθυνση την DG NIR, εξετάζοντας ποιες αντιπροσωπείες είναι πορτοκαλί και κόκκινες. Ε, βλέπουμε και προσωπίες που δεν το περιμέναμε. Για παράδειγμα, η με 79%, 71% σε άλλους τομείς. Η Συρία ήταν και αυτή αναμενόμενη, 69%, πιο χαμηλό επίπεδο από ότι η Υπουργομοδού. Αρμενία 71% και Λίβανος 60% πάνω από 50% δηλαδή των έργων βρίσκονται σε προβληματική, ας το πούμε, φάση. Σημαντικό θα ήταν λοιπόν στο σημείο αυτό να μας πει η Διτζινίρ τι σκοπεύει να κάνει και έχω και κάποιες ερωτήσεις για την Αλβανία. Από την εκθέσει είδαμε ότι στην Αλβανία το ίμιση των υπαλλήλων που φροντίζουν τις συμβάσεις και τους ελέγχου έχει, είχε αλλάξει μέχρι το μέση του 2017. Ήθελα λοιπόν να ενημερωθώ εκ των προτέρων ποια θα είναι η συνέπεια Ποιε θα είναι οι συνέπειε για την Αλβανία αυτή τη τάση. Ύστερα. Προφανώ και χρειάζονται άτομα για τη μετάφραση και στον τομέα τη κοινωνία των πολιτών. Στη Σερβία υπάρχει ένα έργο το οποίο είναι 18% του συνολικού χαρτοφυλακίου, του συνολικού φακέλου, ε, το οποίο είναι κοκκίνο. Δεν έχουμε βρει λύση εδώ και γι' αυτό σημαντικό νομίζω ότι θα αναλάβουμε κάποιε πληροφορίε σε ό,τι αφορά αυτό το μεγάλο για τη Σερβία ε, έργο για την Τουρκία. Πάντα την εξετάζουμε. Φαίνεται ότι δεν αντιμετωπίζει προβλήματα η Τουρκία και είναι μια αντιπροσωπεία προς μίμηση σωστά τα εκτιμώ τα πράγματα ή ε, μήπω υπάρχουν κάποια έντυπα προβλήματα στην Τουρκία. Πάντω πολλά τόσο καλά τα πράγματα παρά όλο, την όλη πολιτική κατάσταση που θα περίμενε κανεί ότι θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά στο θέμα τη ΔΕΦΚΟ. Θα ήθελα να πω το εξή. Ε, εξαιρετική δουλειά και σε ό,τι αφορά η προετοιμασία των στοιχείων ε, πάντα νομίζω ότι κάνει καλή εντύπωση το να δίνουμε στοιχεία τα οποία δεν είναι θετικά γιατί αυτό μας κάνει να έχουμε εμπιστοσύνη στα υπόλοιπα στοιχεία, ξέρετε. Σας ευχαριστώ σε ό,τι αφορά τα προγράμματα χρηματοδότησης τώρα. Δεν μπορούν να εντοπιστούν στο σημείο αυτό. Και έτσι λοιπόν διμερώς θα εκφράσουμε τις επιθυμίες μας και ενδεχομένως να μπορέσουμε να ελέγξουμε καλύτερα τα πράγματα, τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει και τα οποία εντόπισε η ΤΕΦΚΟ πάνω από 10 αντιπροσωπείες που έχουν πάνω από 60% προβληματικά προγράμματα. Σε μία αντιπροσωπεία είναι στο 98% το ποσοστό των προβληματικών project Ερυθρέα, για παράδειγμα. Είναι δύσκολα τα πράγματα σε αυτές τις χώρες, αλλά τι κάνετε πραγματικά για να βελτιώσουμε την κατάσταση, γιατί είναι σχεδόν 100% το 98% καταλαβαίνετε. Τι πώς επικεντρωνόμαστε σε αυτές τις αντιπροσωπείες. Ε, τώρα, δημοσιονομικός, ε, δημοσιονομική υποστηρίξη, σημαντικό το σημείο της EMI. Α, 10 από τα 15 λοιπόν έργα. Τα μεγαλύτερα λοιπόν από αυτά τα project είναι προβληματικά. Κυρίως ε, για θέματα χρηματοδότησης προϋπολογισμού και 8 από τα 15 προγράμματα έχουν να κάνουν με υποστήριξη χρηματοδότησης. Τι έχει γίνει λοιπόν στην υποστήριξη χρηματοδότησης που υπάρχει ουσιαστικά επιδείνωση της κατάστασης. Ε? Αλλά χαιρόμαστε που περιγράφεται και την ε, άσχημη κατάσταση που επικρατεί εκεί ε, με αξιοπιστία. Υπάρχει κάποιος, ε, μια μαύρη λίστα μήπως ε, ή συνεχίζουν τα πράγματα όσο έχουν. Και στη συνέχεια για το KPI 2021 2023 θα λάβω το εξής και τότε στις 10 αντιπροσωπείες ε, με το μεγαλύτερο αριθμό εκκρεμών ελεγχών. Μαγάτα σκάρι εισηγητέλα για τις αυτές τις 10 χειρότερες αντιπροσωπείες. Και έχουν πραγματικά μεγάλη καθυστέρηση σε ό,τι αφορά τους ελέγχους του 2014. Γιατί? Γιατί και τι κάνετε εσείς για να βελτιώσετε την κατάσταση. Κόγκο, Τσάτ και Κεντρική Αφρικανική Δημοκρατία. Δύσκολες χώρες δεν λέω, αλλά και αυτές ε, σημειώνουν αρνητικά αποτελέσματα σε ό,τι αφορά τους ελέγχους. Ποιοι είναι οι λόγοι. Αυτέ τι ερωτήσει είχα να κάνω και δεν ξέρω ποιο θέλει να πάρει το λόγο για να απαντήσει. Ευχαριστώ. Όπω θέλετε. Uh, Madam Chair, you, you... Κυρία Πρόεδρε, αναφέρατε μία σειρά αντιπροσωπιών που έχουν προβλήματα με τα project. Δεν μπορώ να σας κάνω σχόλια για την κάθε μία ξεχωριστά, γιατί δεν έχω μαζί μου όλα αυτά τα στοιχεία σε αυτό το στάδιο. Αυτό που κάναμε ξεκάθαρα όμως ήταν να έχουμε συζητήσει με τις ε, αντιπροσωπείες ε, και να τους ε, δείξουμε ξεκάθαρα την ανάγκη να αναλάβουν άμεση δράση. Ε, θα σημειώσω αυτά που είπατε σχετικά με το που βρισκόμαστε όσον αφορά στην ΔΕΦΚΟ. Φυσικά προσπαθούμε να βαθμονομήσουμε τις ε, ε, προσπάθειές μας βάση των βέλτιστων πρακτικών. Όλη αυτή η φιλοσοφία των KPIs έχει αναπτυχθεί από την DEFCO για να έχουμε περαιτέρω πρόοδους. Η εφαρμογή τους λοιπόν θα μας βοηθήσει να κερδίσουμε το χαμένο χρόνο. Δεν μπορώ να σας εγγυηθώ ότι αυτό θα γίνει αμέσως, αλλά αυτό είναι ο στόχος. Αναφέρατε ε, την Τουρκία, έχουμε προβλήματα, έχουμε προκλήσεις. Μία από αυτές είναι η εφαρμογή των προγραμμάτων. Έχουμε ε, πολλά από θέματα που ακόμα δεν έχουν ρευστοποιηθεί, όμως η κατάσταση στην Τουρκία είναι τελείως διαφορετική από ό,τι είναι στις άλλες χώρες, γιατί εκεί έχουμε εφαρμογή από την χώρα δικαιούχο, δηλαδή τη διαχείριση την έχουν οι τουρκικές αρχές. Άρα η άσκηση των φαναριών εκεί δεν γίνεται με τον ίδιο τρόπο. Έχουμε αυτές τις προκλήσεις, τις αντιμετωπίζουμε και κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν να διασφαλίσουμε ότι οι τουρκικές αρχές θα επιταχύνουν την εφαρμογή των προγραμμάτων. Όμως ξέρετε πως η κατάσταση στην Τουρκία αυτή τη στιγμή είναι ιδιαίτερα προβληματική. Υπάρχουν διάφοροι παράγοντες που επηρεάζουν, θα έλεγα, την κατάσταση. Και είναι δύσκολο να διαχειριστούμε το τι συμβαίνει. Και φυσικά έχουμε και τη διευκόλυνση για τους πρόσφυγες, η οποία ξεκίνησε πέρυσι να εφαρμόζεται και η οποία θα μπει στα νούμερα του 2017 για να μας δείξει μια καλύτερη εικόνα από ό,τι είχαμε το 2016. Για τις αλλαγές προσωπικού στην Αλβανία, δυστυχώς Αυτές οι αλλαγές προσωπικού είναι ένα από τα προβλήματα με τα οποία ερχόμαστε αντιμέτωποι στις αντιπροσωπείες και απλώς πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε και να λάβουμε μέτρα για να περιορίσουμε τις επιπτώσεις στην εφαρμογή των προγραμμάτων. Και φυσικά υπάρχουν κάποια σημαντικά προγράμματα που αυτή τη στιγμή εφαρμόζονται ε, στην Αλβανία. Έχουμε ε, ε, μεγάλο πολιτικό κεφάλαιο εκεί στην Αλβανία. Η έχει μεγάλη δουλειά να κάνει λόγω της διεύρυνσης. Δεν έχουμε βέβαια ε, πρόβλημα διότι ο επικεφαλής της αντιπροσωπείας εκεί είναι πολύ ικανός και το προσωπικό που ήρθε, το καινούριο προσωπικό είναι ιδιαίτερα ικανό και αυτό άρα ε, δεν θα έχουμε μεγάλες ε, αποκλήσεις από αυτή την αλλαγή προσωπικού που είναι κάτι αναπόφευκτο. Τώρα για τη Σερβία. Ίσως ε, επανέλθω όταν θα τα δω λίγο πιο λεπτομέρως εδώ στις σημειώσεις μου γιατί είναι μία από τις χώρες που πραγματικά δεν έχω στο μυαλό μου έτσι απλά. Να δώσω λίγο το λόγο στο Λουκ για να μιλήσει και αυτός για τις δικές του. Περιμένουμε τις πληροφορίες για τη Σερβία γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία για την απαλλαγή ε, γραπτός αν μπορείτε. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Αναφέρουμε στην έκθεσή μας εννέα αντιπροσωπείες στις οποίες δεν έχουμε επιτύχει τους στόχους σε επίπεδο KPIs. Αυτές φυσικά έχουν μετρήσεις ε, επιδόσεων ε, για όλους τους KPI, τους 24 δηλαδή KPIs, όχι μόνο τους δύο που ε, είναι στο project φανάρι, κόκκινο, πράσινο, πορτοκαλί. Η Επίτροπη Μίμητσα και αν ξέρουν αυτά τα στοιχεία, υπάρχει πιο συγκεκριμένη ανάλυση για αυτούς τους KPIs και υπάρχουν και οι 10 αντιπροσωπείες οι οποίες που έχουν το πιο μεγάλο ποσοστό στο φάκελο των κόκκινων και των πορτοκαλί project. Έχουμε λοιπόν μια άλλη λίστα η οποία ξεκινά με την Ιεμένη, Ερυθρέα, Μποσουάνα, Μαλή, Βοζαμβίκη, ε, Μαυριτανία, Λεσόθ, Λέσοθο, Μεξικό και το Νότιο Σουδάν. Για να δείτε λίγο το έβρος ε, του φακέλου αυτού. Σε αυτές τις περιπτώσεις, όπως και σε όλους τους άλλους KPIs, ζητάμε από την Γεωγραφική Διεύθυνση και από την Αντιπροσωπεία να φτιάξει ένα σχέδιο δράσης, κατά περίπτωση και ανάλογα με τα αίτια που εντοπίζονται. Και για αυτούς τους δύο KPIs λοιπόν και για τις υπόλοιπους η αντιπροσωπεία θα πρέπει να μπορεί να είναι σε θέση, δηλαδή να μας πει ποια είναι τα μέτρα που θα βελτιώσουν την κατάσταση. Και αυτό όχι μόνο για να μπορέσουμε να μιλήσουμε στο Συμβούλιο και στο Κοινοβούλιο και να εξηγήσουμε ε, γιατί, ότι πήγαν πίσω οι KPIs, αλλά για να μπορέσουμε να δείξουμε και ένα ε, σχέδιο δράσης. Εδώ είναι σημαντικό να προσέξουμε πώς ερμηνεύουμε τους KPIs και τα διάφορα χρώματα που δίνουμε στα project. Το να σταματά ένα project ή να αναστέλλεται η δημοσιονομική υποστήριξη ή να καθυστερείται η καταβολή μιας δόσης επειδή δεν πληρούνται οι όροι, ε, σημαίνει ότι είτε θα πάρει ε, πορτοκαλί είτε κόκκινο χρώμα το project, όμως τα χρήματα δεν έχουν δοθεί. Δεν κατεβλήθηκαν τα χρήματα, υπήρξαν καθυστερήσεις στην εφαρμογή του project, άρα θεωρούμε πως μπορεί να μπει στα κόκκινα και επειδή δεν δίνουμε τα χρήματα και μετά υπάρχουν οι καθυστερήσεις, θεωρούμε ότι είναι δύσκολο, αλλά όχι αδύνατο ξανά ε, ξεκινήσει η συνεργασία να πετύχουμε τους στόχους. Όμως τα χρήματα δεν έχουν δοθεί, δηλαδή έχουμε προστατέψει τα χρήματα των φορολογουμένων. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να γνωρίζετε ότι στα πλαίσια της δημοσιονομικής υποστήριξης οι καθυστερήσεις καταβολής επειδή δεν πληρούνται οι όροι είναι αυτές που δίνουν την κόκκινη ή πορτοκαλί σημαία στα προγράμματα. Και ε, μπορεί με να φαίνεται στους καταλόγους ε, το ποσό ε, γιατί είναι τα πιο σημαντικά project αυτά και εμφανίζονται στα top 10 των project. Τώρα, για την εφαρμογή των εξωτερικών ελέγχων. Υπάρχουν εξωτερικοί έλεγχοι που έχουν ένα πλάνο σε τρία, που διαρκεί τρία χρόνια και έχουμε έλεγχο κάθε χρόνο. Συνήθως όταν έχουμε καθυστέρηση στους εξωτερικούς ελέγχους έχουμε και καθυστέρηση στην συνεργασία γιατί επειδή δεν υπήρξαν συμβόλαια δεν υπήρξαν και εξωτερικοί έλεγχοι και επειδή συνήθως η συνεργασία είναι περίπλοκη το ίδιο γίνεται και με τους εξωτερικούς ελέγχους οι προθεσμίες είναι πιο μεγάλες, πιο μακρινές. Ε, γενικά η περίοδος ε, προβληματικών ε, συναλλαγών και ανταλλαγών είναι περί πιο μεγάλη. Άρα και το planning, ο σχεδιασμός δεν είναι ρεαλιστικός. Όταν μιλάμε λοιπόν για χρηστή δημοσιονομική διαχείριση θα πρέπει σε βραχυπρόθεσμο επίπεδο να έχουμε ρεαλιστικά σχέδια, να έχουμε την πιο λεπτομερή αξιολόγηση και την πιο σωστή ε, αξιολόγηση των δυνατότητας να τηρήσουμε το σχέδιο και μετά να δούμε λίγο και ποιο είναι ο λόγος που συμβαίνουν όλα αυτά. Δεν υπάρχει προσωπικό, δεν υπάρχει κατάρτιση στο προσωπικό. Και στο τέλος φυσικά να δούμε και τα μέτρα που θα μας βοηθήσουν να βελτιώσουμε την κατάσταση για το σύνολο των KPIs. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ για τις πολύ σημαντικές απαντήσεις που ξεκαθαρίζουν τα πράγματα. Να πω όμως ότι ε, θα πρέπει να ξέρουμε και πώς οι, ε, οι πρέσβεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης θέλουν να αντιμετωπίσουν το θέμα. Ποιος είναι αυτός που υπογράφει. Είναι πρόβλημα του ανωτέρου, του ε, κατωτέρων. Θα ε, υπάρχει κάποια διπλωματική διάσταση σε αυτό το θέμα. Ε, και από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι σημαντικό αυτό και σε οικονομικό επίπεδο. Θα θέλαμε λίγο να μας πείτε κάποια πράγματα για αυτά. Α, και ε, να ακούσαμε ότι η, κάποια μέλη της αντιπροσωπείας του Αφγανιστάν ασχολούνται με το εμπόριο του αλκοόλ. Τα διάβασα στην εφημερίδα. Είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε ποιοι είναι αυτοί. Είναι συνεργάτες της Κομισιόν, είναι άτομα της Κομισιόν ή είναι ντόπιοι. Παρακαλώ. Ε, για τον ε, πρέσβη πρώτα και μετά για την άλλη ερώτηση. Να πω ότι Είμαι αρκετά ικανοποιημένο με τον τρόπο που οι πρέσβει ανταποκρίθηκαν γιατί νομίζω ότι υπάρχει όλο και περισσότερη κατανόηση και μέσα στον χρόνο βελτιώνεται η κατάσταση ούτω ώστε να εξασφαλίζεται το ότι όλα θα γίνονται όσο καλά μπορεί να γίνουν και πάρα πολλέ φορές με δύσκολες συνθήκε Εμεί ε, δεν ε, ε, διστάζουμε έτσι κι αλλιώ οι εκθέσει υποβάλλονται από τους ε, πρέσβει και πιστεύω ότι αυτέ οι εκθέσει είναι ένα πάρα πολύ χρήσιμο εργαλείο γιατί έτσι μπορούμε να καθορίσουμε τι αρμοδιότητε κάστου, τι ευθύνε εκάστου. Επισημαίνουμε ότι πρέπει, υπάρχει έτσι επομένω ε, η συνειδητοποίηση. Ε, κινητοποιούμε τους πρέσβες ε, όποτε και όταν χρειάζεται και επίσης σε τακτά διαστήματα τα συζητούμε οπότε και κάποια στιγμή αρχές του χρόνου πρόκειται να υπάρξει κάποια συνάντηση αρχάς του έτους για να τα ξαναπούμε και για να ξανατονίσουμε ε, όπως πάντα γίνεται σε αυτές τις συναντήσεις ότι πρόκειται για κάτι που δεν είναι καθόλου αφηρημένο αλλά το ότι αυτό είναι μια διαδικασία λογοδοσίας ε, κοινοβουλευτικού ελέγχου του Κοινοβουλίου επί της Επιτροπής. Η Πρόεδρος. Όχι, συγγνώμη. Ο κύριος Όσον αφορά τους πρέσβες, νομίζω ότι πέρασε κάποια περίοδος προσαρμογής μετά από την συγκρότηση αυτής της ε, Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης. Ε, αυτοί, κάποιοι προχωρούσαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ε, και οι πρέσβες από τα κρατημέλη όμως δεν ξέρανε όπως οι προερχόμενοι από την Επιτροπή τα, τα σχετικά με τον προϋπολογισμό και τα της διαχείρισης, κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό όσον αφορά το χαρτοφυλάκιο κάποιας ε, ε, αντιπροσωπείας, γιατί 70% ε, της δουλειάς της αντιπροσωπείας είναι συνεργασία, άρα πολύ σημαντικός τομέας και ξέρουν επικεφαλής ότι έχουν την ευθύνη και την αρμοδιότητα και τι γίνεται με τη σχετική δήλωση αξιοπιστίας στα τέλη κάθε χρήσης οπότε ε, εμείς αναλύουμε ε, κάθε τέτοια έκθεση και καταρτίζεται ένα πρόγραμμα δράσης, δεσμεύονται την προσωπία σε αυτού και έτσι διορθώνεται ε, η ρότα <coughs> των ε, αντιπροσωπιών και συζητούμε σε ψηλό επίπεδο τα των επιδόσεων ε, όσον αφορά κάθε γεωγραφική ζώνη και επίσης και γίνονται κάποια περιφερειακά συνέδρια και εκεί πηγαίνουν επικεφαλής συζητείται ο προγραμματισμός ελέγχονται το ποια είναι τα προγράμματα και λοιπά Οπότε έτσι έχουμε εξέταση όλων των ε, προβλημάτων, όλων των δικτών που δεν είναι στα επίπεδα που θέλουμε. Βεβαίω ε, υπάρχουν ε, διαφορετικές κουλτούρες, διαφορετικές παραδόσεις σε κάθε χώρα και, σε, έτσι έχει διαφορετική κουλτούρα ο κάθε πρέσβης, αλλά τελικά έχουμε αυτή τη συνεργασία και εσείς άλλωστε τους τα τονίζετε για να ταξιδεύετε το Αφγανιστάν τώρα. Δεν έχω δυστυχώ τα στοιχεία. Εντάξει, έγινε αυτή η διαρροή στον τύπο για α, το αλκοόλ, το ενόπνευμα τέλο πάντων σε αντιπροσωπεία. Καλά, καλά, θα σας στείλω. Θα σας στείλω τα μέσα ενημέρωση τα σχετικά, λέει ο Πρόεδρος. Πριν από τρεις-τέσσερις ε, μέρες διαβάσαμε. Όλες τις λεπτομέρειες. Ε, γι' αυτό σα τα έλεγα, λέει η κυρία Γκρέσλε. Τώρα, για να δούμε επόμενε φάσεις για τα EAMR. Το benchmark για τους ε, δείκτες ε, είναι 60%. Εσεί πώς θα συνεχίσετε με αυτό το 60%? Φτάσαμε στην οροφή ή όχι. Πώς θα εξεταστεί η υπόθεση των εκθέσεων τα επόμενα χρόνια. Μπαζέ. Ο στόχο είναι να έχουμε 100% στο πράσινο για όλε τι Αλλά δεν μπορεί να είναι όλα τέλεια και οπότε έχουμε αυτό το 60% ως κατόφλι γιατί από το κατόφλι αυτό ε, έχουμε ένα πρόγραμμα για βελτίωση της κατάστασης. Αυτό δεν σημαίνει ότι αναδείκτη ακόμα και πάνω από το 60% εάν δεν πετύχουμε το KPI ότι δεν πρέπει να κάνουμε ό,τι χρειάζεται για να πετύχουμε το στόχο. Ο στόχος είναι για τις 9 αντιπροσωπείες κατά το 60% ή πάνω από το 60% να υπάρχει πρόοδος για όλες τις αντιπροσωπείες και επίσης σας παραλαμβάνω, αν όχι το 18, για το 19 και για το 20 πρόκειται να αλλάξουμε κάποιους δείκτες και θα εστιαστούμε σε άλλες προβληματικές και ίσως να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε από πιο κάτω για να προοδεύσουμε κάποιες αντιπροσωπείες σε κάποια μέτωπα τα οποία τώρα παίζονται και διακυβεύονται. Συμφωνώ, συμφωνώ με τον ε, Λιουκ. Ε, έχουμε αυτό το 60% για τα KPIs που είναι το benchmark. Ε, θα πρέπει το 60% τουλάχιστον να επιτευχθεί. Να, να, αυτό είναι το, βασικό. αυτό όμως δεν είναι ε, Όπως η, η διαφάνεια που έδειξα πριν, που δείχνει ότι υπάρχουν κάποιες αντιπροσωπίες οι οποίες ε, πάνε πάνω από το 90% στους δείκτες. Ο στόχος μας λοιπόν είναι να αυξήσουμε το επίπεδο όλων, αλλά ταυτόχρονα επειδή υπάρχει και το κίνητρο εδώ, να μην θέτουμε και στόχους οι οποίοι δεν είναι εφικτοί σε κάποιες περιπτώσεις. Πρέπει λοιπόν να, διαβάζουμε, να λαμβάνουμε υπόψη ότι σε κάποιες περιπτώσεις είναι πολύ δύσκολο για κάποιες αντιπροσωπείες να ξεπεράσουν το 60%. Σε άλλες περιπτώσεις όμως όπου υπάρχει ένα φυσιολογικό περιβάλλον όπως θα λέγαμε αν οι επιδόσεις είναι στο 60% θέτουμε ερωτήματα. Και αυτά είναι και τα στοιχεία που στέλνουμε και στις αντιπροσωπείες. Να επανέλθω λίγο στο προηγούμενο ερώτημα για τους πρέσβεις, γιατί ε, κάτι άλλο σκέφτομαι. Ε, συγκεκριμένα για τις περιοχές ε, της διεύρυνσης αλλά και για τις περιοχές γειτονίας ένα από τα πράγματα που μας βοήθησαν στο να κάνουμε λίγο πιο υπεύθυνου τους επικεφαλείς των αντιπροσωπιών είναι ότι τώρα υπάρχει πραγματική κατανόηση πλέον ότι η εξωτερική βοήθεια, τα χρήματα που δίνουμε σε αυτές τις τρίτες χώρες είναι ένα ιδιαίτερα σημαντικό εργαλείο στις σχέσεις μας με αυτές τις τρίτες χώρες. Μπορούμε να μοχλεύσουμε και ακριβώς αυτό προσπαθούμε να κάνουμε κινητοποιήσουμε ε, ως προς τις αλλαγές που πρέπει να γίνουν, γιατί οι αλλαγές που θα γίνουν εκεί είναι καλές και για εμάς. Με αυτή τη συνειδητοποίηση λοιπόν υπήρξε περισσότερη κατανόηση και επικέντρωση στη βοήθεια ε, για να χρησιμοποιηθεί με το σωστό τρόπο. Ο συνάδελφος, ε, η συνάδελφος Σμίτ παρακαλώ. Ναι, ευχαριστώ. Να πω κάτι ε, που είναι πολύ σημαντικό γιατί δεν έχω καταλάβει ε, αυτή την κατανομή ε, βοήθεια στον δημοσιονομικό επίπεδο και για τα καλά και για τα κακά project. Δεν το έχω καταλάβει καλά. Και μιλάτε συνέχεια για αυτά τα προβληματικά project. Το 1 τέταρτο αυτό είναι προβληματικά εντός εισαγωγικών. Δηλαδή, είπατε βέβαια ότι τα χρήματα δεν έχουν δοθεί. Τι δείχνει, ε, τι ορίζεται ως προβληματικό. Αναφέρατε πάρα πολλές φορές επίσης ότι κάνετε τακτικές συζητήσεις σε δικό σας επίπεδο και σε όλα τα επίπεδα. Κατά την άποψή μου όμως οι συζητήσεις δεν λύνουν τα προβλήματα. Ε, είπατε μετά ότι θέτετε ερωτήματα. Ε, εντάξει, καλά να θέτουμε ερωτήματα, αλλά να έρχεται και η απάντηση. Ποιος είναι ο στόχος σας. Ο στόχος ε, θα πρέπει να είναι να φτάσουμε στο 100%. Δεν ικανοποιού, ε, δεν μπορούμε να λέμε ότι ικανοποιούμαστε με λιγότερα γιατί όλα είναι τόσο δύσκολα. Είναι δύσκολες αυτές οι χώρες ούτως ή άλλως. Εμείς όμως θα πρέπει να προσπαθούμε να χορέψουμε όπως πάνω σε αυγά οι πρέσβεις ε, λένε εντάξει καλά πάνε τα πράγματα, οι άλλοι λένε παρόλα αυτά υπάρχει πρόβλημα, η αντιπροσωπεία είναι και έτσι και αλλιώς, αλλά γίνουμε λίγο πιο ξεκάθαροι. Παρά λοιπόν τα αποτελέσματα θα ήθελα να είμαστε λίγο πιο συγκεκριμένοι και να είμαστε λίγο περισσότερο αφιερωμένη στο στόχο μας ε, γιατί πρόκειται πραγματικά για χρήματα φορολογουμένων και δεν θα έπρεπε να είμαστε έτσι χαλάροι. Κατά την άποψή μου, ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση πιο πολλοί ερωτήσει τίθενται παρά απαντήσεις δίνονται, αλλά ας απαντήσουν και οι υπεύθυνοι, παρακαλώ. Κοιτάξτε, για την δημοσιονομική υποστήριξη αν θέλετε, θα απαντήσω. Έχουμε δύο KPIs που έχουν ως στόχο να μετρήσουν δύο συγκεκριμένες καταστάσεις. Πρώτον, το αν ένα ε, ε, project, ένα έργο έχει καθυστέρηση. Για παράδειγμα, πρέπει να εκταμιεύσω ένα συγκεκριμένο ποσό σε σχέση με κάποιους στόχους που έχουν τεθεί ε, το πρώτο έτος και το δεύτερο έτος έχω ένα δεύτερο κομμάτι της χρηματοδότησης σύμφωνα με άλλους στόχους. Και μετά έχω έναν άλλο δείκτη, ο οποίος μετρά την δική μας αξιολόγηση της δυνατότητας που έχουμε να επιτύχουμε το στόχο. Μπορεί να μετρηθεί λοιπόν σε τριετές ε, ε, διάστημα ο στόχος συνολικά, όμως σε αυτή τη φάση που βρισκόμαστε είμαστε σε θέση να επιτύχουμε τελικά το στόχο στην τριετία. Όσον αφορά λοιπόν στη δημοσιονομική υποστήριξη, η οποία μπλοκάρεται επειδή δεν τηρούνται οι προϋποθέσεις. Και, για... και στην ε, περίπτωση αυτή φυσικά ε, δεν μπορώ να εκταμιεύσω, να καταβάλω χρήματα. Ε, έχω καθυστέρηση. Είναι προβληματικό λοιπόν το ε, project. Είναι κόκκινο. Ακόμα και αν δεν έχω καταβάλει χρήματα και δεν έχω κάνει την εκταμείευση. Απ' την άλλη βέβαια, αν δεν δώσω τα χρήματα, στα τρία χρόνια δεν θα πετύχω τους στόχους. Ακόμα και αν εγώ έχω κρατήσει τα χρήματά μου. Και γι' αυτό το λόγο είναι κόκκινα τα project. Πρέπει λοιπόν να διαχωρίσουμε το γεγονό ότι είναι στα κόκκινα ένα project από τι επιπτώσει. Το ότι είναι στα κόκκινα δεν σημαίνει ότι θα έχει δημοσιονομικέ επιπτώσει. Στη δική μα περίπτωση δεν θα έχει. Αλλά αν ένα project παραμείνει στα κόκκινα, οι δικοί μας στόχοι σε επίπεδο ανάπτυξης δεν έχουν επιτευχθεί. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Έτσι λοιπόν αυτό που είχαμε προβλέψει για τους εταίρους μας δεν επετεύχθη. Ακόμα λοιπόν και αν δεν δοθούν τα χρήματα, το project είναι στα κόκκινα γιατί υπάρχει πραγματική δυνατό, ε, δυσκολία να επιτύχουμε τους στόχους μας και φυσικά να δώσουμε τα χρήματα. No, I, ε, Βέβαια και συμφωνώ με όλα όσα ε, είπε ο Πολύ ε, καλή ανάλυση του πώς έχουν τα πράγματα και να το ξεκαθαρίσουμε ότι υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις, ίσως κάποιο πρόγραμμα το οποίο είναι στην φάση της σύλληψής του. Και αυτό είπα προηγουμένως όταν συζητούσαμε για τους δείκτες, ότι τότε σε εκείνη τη φάση λοιπόν υπήρχαν ερωτηματικά όσον αφορά τη λογική της παρέμβασης, οπότε σε κάποιες ε, φάσεις έχουμε επιδείξει υπερβολική φιλοδοξία. Άρα αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να δούμε πώς θα κάνουμε ε, τη διάκριση μεταξύ της ε, συμβολής και της επιδίκασης. Οπότε ε, να έχουμε ένα στόχο, να έχει σχέση με την παρέμβαση ή από την άλλη μεριά να έχουμε ένα στόχο που να βοηθά στην ε, επίτευξη του στόχου. Ε, και από την άλλη μεριά είμαστε υπερόπτες, είμαστε υπερβολικά φιλόδοξοι και γι' αυτό να γίνεται αυτή η διάκριση, οπότε και να μπορούμε να συγκροτήσουμε ένα πρόγραμμα το οποίο να επιδέχεται επαναξιολόγηση των δυνατοτήτων του τι μπορούμε να κάνουμε και τονίζουμε επίσης ότι με αυτό το σύστημα των φαναριών ε, έχουμε κάποια υγιή διαχείριση του χαρτοφυλακίου και υποψιάζουμε ότι ακριβώς το ίδιο σύστημα έχουν πολλές επιχείρησεις. Αυτό καθορίζει το πώς θα γίνει η διαχείριση της εταιρείας Οπότε για τα φανάρια εξαρτάται ποιο δίκτυ κάθε φορά μετερχόμαστε για να μπορέσουμε να καταγράψουμε την πραγματικότητα, να δούμε αν υπάρχει καθυστέρηση, αν ενεδρεύει κάποιος κίνδυνος για το στόχο κλπ. Όμως κάποιες φορές αυτά ε, πηγάζουν από δικό μας λάθος, αν έχουμε επιδείξει υπερβολική φιλοδοξία. Πολλές φορές όμως φταίνε ε, άλλοι εξωτερικοί παράγοντες. Να, παράδειγμα, δημοσιονομική στήριξη ε, στην Γενική Διεύθυνση ΝΙΡ. Να είπαμε και για την ε, ε, Ουκρανία που προσφέρουμε τη υποστήριξη και εκεί υπάρχει θεσιμότητα που αφορά την εκπλήρωση κάποιων νομοθετικών υποχρεώσεων. Αν όμως δεν έχει πιστεί αυτή η νομοθεσία, εμείς δεν θα εκταμιεύσουμε αυτά τα οποία πρέπει. Ε, να την παναπεί σωστή στη διαχείριση, να την παναπεί μόχληση. Ε, οπότε, αν δεν γίνει εκταμίευση τη μια χρονιά, δεν γίνονται την επόμενη και δεν θα γίνει ε, ε, άπαξ και δεν πληρούνται σχετικές προϋποθέσεις όμως πέραν όλων αυτών των παραγόντων υπάρχουν και άλλες μεταβλητές. Να, ας πούμε, η στήριξη της κοινωνίας των πολιτών μέσα σε μια δύσκολη συγκυρία, κάτι το οποίο συμβαίνει συχνά στη δουλειά μας. Οπότε όσοι καλύτερες και να έχει κάποιος, ε, θα πρέπει να ληφθεί η απόφαση για κάποιο πρόγραμμα επί ε, Μπορεί να υπάρχει κόκκινο φανάρι. Αναγνώριση κάποιων φορέων κοινωνίας πολιτών, αλλά αυτό το οποίο κάνουμε είναι δυναμικά ε, τη λύση, τον τρόπο να παρακάμψουν αυτές τις δυσκολίες. Θα ήθελα να ευχαριστήσω για την εξήγηση του συστήματος με τα φανάρια ε, ε ευχαριστώ, το κατάλαβα. Δεν είμαι φίλος ε, της ε, ενίσχυση αυτής ε, ενίσχυσης και υποστήριξης. Δεν καταλαβαίνω γιατί κάθε χρόνο το χειροκροτάμε, αλλά πρέπει να σας πω ότι πραγματικά εσάς σας βρίσκω εξαιρετικού και η ισοδοξία σα είναι εξαιρετική, αλλά φαντάζομαι ότι οι στόχοι αυτοί καθορίζονται από εμπειρογνώμονε. Ένα τέταρτο των, των έργων είναι προβληματικά. Θα ήθελα λοιπόν να το εξετάσουμε αυτό, να είναι πιο ρεαλιστική η στόχη. Δεν είναι δυνατόν να μην ξέρουν αυτοί που καθορίζουν τους στόχους, πω έχει η κατάσταση επιτόπου. Άρα, Καλή και αισιοδοξία, συγχαρητήρια. Άρα θεωρώ ότι αν ένα στα τέσσερα προγράμματα παρουσιάζει πρόβλημα, είναι μεγάλο ποσοστό η πρόεδρο. Κοιτάξτε, το ένα τέταρτο των έργων είναι προβληματικά. Το ότι το γνωρίζουμε αυτό είναι ήδη μια πρόοδο. Κανεί δεν θέλει να μείνει σε αυτό το επίπεδο φυσικά το ποσοστό αποτυχία και προφανώς όλοι ανησυχούμε όταν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Έχουμε την εντύπωση ότι τουλάχιστον το γεγονός ότι σημειώνουμε αυτά τα ποσοστά είναι θετικό. Σας ευχαριστώ. Δεν θεωρούμε ότι υπάρχει κάποια απειλή. Μια υπόσχεση τα λέγαμε, μάλλον, για περαιτέρω ανάλυση της, ε, των αναφορών αυτών. Και πραγματικά αυτό γίνεται από τις Γενικές Διευθύνσεις και εγώ προέβησα σε ανάλυση των εκθέσεων, εξεταστά και τα στατιστικά στοιχεία. Σας ευχαριστώ λοιπόν και ε, σας καλώ να παρακολουθούμε συνέχεια το θέμα αυτό γιατί εκεί νομίζω ότι δεν υπάρχει οποιοδήποτε κίνδυνος αν συνεχίσουμε να παρακολουθούμε το θέμα αυτό. Είναι σημαντικό λοιπόν να είναι σε διαρκή επαγρύπνηση οι αντιπροσωπείες για να πετύχουν καλύτερα αποτελέσματα. Και νομίζω ότι το benchmark του 60% σας κατανοούμε, σας καταλαβαίνουμε. Αλλά νομίζω ότι μπορούμε να βελτιώσουμε και το άνω περιθώριο. Σας ευχαριστώ πολύ και για την εργασία σας. Σας ευχαριστώ πολύ γιατί είναι πραγματικά εξαιρετική. Και έτσι ολοκληρώσαμε το θέμα αυτό και περνάμε στο σημείο 8 για την πολιτική για τα κτίρια στο Λουξεμβούργο. Και να σας καλωσορίσω, ε, κυρία Χόλμαϊρ, που είναι από την Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού η υπεύθυνη για τα κτίρια αυτά. Σας καλωσορίζω. The head of OEL. Yeah, thanks, thanks for coming. Welcome. Σας ευχαριστώ που ήρθατε και καλώς ορίσατε. Και η κυρία Χόλμα ήρθε να πάρει το λόγο για ένα ασυνήθιστο project το οποίο θέλει να μας παρουσιάσει σήμερα. Αγαπητοί Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, δεν θέλω να παρουσιάσω όλο το project, αλλά να σας ε, αναφέρω τι μου έκανε εντύπωση σε ό,τι αφορά τα κτίρια, σε ό,τι αφορά το κτίριο Ντρόσμπαχ ε, και τη δεύτερη πτέρυγα. Στο Λουξεμβούργο, λοιπόν, στην παρούσα φάση, νοικιάζουμε κτίρια με αποθήκες, με χώρους εργασίας. Μας οδήγησαν αυτά και σκέψεις για την προστασία. Δεν ε, μπορέσαμε λοιπόν να βρούμε ένα σωστό κτίριο στο Λουξεμβούργο, το οποίο θα το χρησιμοποιούσαμε ως αποθήκη και ως ε, ε, χώρο εργασία. και έτσι λοιπόν καταλήξαμε στο κτίριο Ντρόσπακ, το οποίο δεν είναι ενδεχομένω το πλέον ενδεδειγμένο για τις εργασίες αυτές, αλλά δεν υπήρχε την εναλλακτική. Είχαμε και τα θέματα ασφάλειας και τα θέματα πυροπροστασία. Τα λάβαμε όλα αυτά υπόψη. Κοιτάξαμε και την διάτρωση του κτηρίου και είδαμε κάποια συνήθιστα στοιχεία, τα οποία ενδεχομένω σήμερα, έτσι, ε, ναι, 2017, δεν είναι σύγχρονα. Για παράδειγμα, το γεγονός ότι είχαμε από θέματα και καφέ και τροφίμων αποθηκευμένα. Αν ρωτιέμαι γιατί αποθηκεύονται έτσι, γιατί οι καθημερινές ανάγκες για να καλύπτονται δεν χρειάζεται να υπάρχει τέτοια μεγάλη αποθήκευση τόσο μεγάλο αποθέματο. Νομίζω ότι σήμερα, τη σημερινή μέρα αυτά τα παραδείγματα τελευταία στιγμή, just in time, ε, ανάλογα με τι ανάγκε. Και για παράδειγμα στα τυπογραφία. Να πω ότι δεν υπάρχει συνεργασία μεταξύ των ε, θεσμικών οργάνων. Ε, γιατί κάνουν τι εκτυπώσεις του ξεχωριστά όλα τα θεσμικά όργανα, χωρί καμία συνεργασία. Και έτσι λοιπόν προκύπτουν διάφορες τέτοιες ε, ιδιαιτερότητες και ρωτώντας διαπιστώσαμε το πώς γίνεται η αποθήκευση, η διανομή, η εκτύπωση και ότι όλα αυτά δεν ε, είναι σύγχρονα. Χρειάζεται ανανέωση των ε, διαδικασιών. Δεν είχαμε και χρόνο φυσικά, υπήρξε μεγάλη χρονική πίεση. Ε, νομίζω ότι χρειάζεται σίγουρα συνεργασία και μεταξύ των θεσμικών οργάνων. Δεν είναι μόνο το θέμα του Κοινοβουλίου, είναι και το δικαστήριο, είναι και το ελεκτικό συνέδριο. Έχουμε και κτίρια τη Επιτροπή. Ε, έχουμε πολλά μαζεμένα θεσμικά όργανα, για παράδειγμα, σε ό,τι αφορά τα τυπογραφία. Δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να έχει ξεχωριστό τυπογραφείο κάθε θεσμικό όργανο, γιατί να μην υπάρχει συνεργασία και σε ό,τι αφορά την αποθήκευση. Αναρωτιέμαι γιατί αποθηκεύονται τόσο, μεγάλα, τόσο μεγάλες ποσότητες. Ε? Γιατί συνήθω οι πληροφορίες που μας έδιναν είναι ότι πρόκειται για μακροπρόθεσμες ε, αποθηκεύσεις. Δηλαδή πράγματα τα οποία μένουν ολόκληρους μήνες στις αποθήκες. Ε. Αυτό γίνεται στη δεκαετία του 70. Μάλιστα, τότε. Είχαμε αλεύρια, καφέ, ρύζι στις αποθήκες. Σήμερα όμως δεν ήθιστε αυτό. Ούτε στον καφέ, ούτε στο τσάι. Υπάρχουν συστήματα επιμελητίας τα οποία τελευταία στιγμή, βράχει πρόθεσμα, κάνουν παραδόσεις. Και τίθεται και θέμα outsourcing. Κατά πόσον ε, είναι θέμα το οποίο πρέπει να το φροντίζει κάθε θεσμικό όργανο από μόνο του. Μήπω θα πρέπει να το αναθέσει αυτό εξωτερικά σε κάποια υπηρεσία. Δεν είχαμε χρόνο να κάνουμε τέτοια ανάλυση. Σε μια γνωμοδότηση όμω ζητούμε να κοιτάξουμε λίγο το θέμα της ε, διάρθρωσης ε, της οργάνωσης. Είχαμε και μία γραμματοδότηση στο παρελθόν, ε, όπου είχαμε ζητήσει να αφήσουμε το σύντομα το, το κτίριο Ντρόσπαχ και να επιστρέψουμε στα βασικά κτίρια. Το κόστος φυσικά θα είναι υψηλό. Αναφέρθηκε ότι δεν υπάρχουν πολλά κτίρια στο Λουξεμβούργο. Ναι, αλλά άμα δεν υπάρχουν αρκετά κτίρια, μήπως θα πρέπει να βγούμε και λίγο εκτός Λουξεμβούργου. Να βρούμε τρόπους άλλους, ε, εφόσον δεν υπάρχουν επαρκή κτίρια. Το κόστος τώρα, σύμφωνα με τις τρέχουσες εκτιμήσεις, δεν είναι και αμεληταίο. Γιατί μιλάμε για συνολικό κόστος αυτής της μεταβατικής λύσης και του κόστους ε, λειτουργίας και ε, συντήρησης είναι 1,7 εκατομμύρια το χρόνο. Ε, δεν είναι για χώρους αποθήκευσης αμαγικά το ποσό, σε καμία περίπτωση. Γι' αυτό όλοι ζητώ και από την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού να ελέγξουν αυτές τις αλλαγές ό,τι αφορά τους χώρους αποθήκευσης και εργασίας, να αλλάξει λίγο ο τρόπος λειτουργίας, να προσαρμοστεί στις σύγχρονους καιρούς, εν πάση περιπτώσει. Σας ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τι θα κάνει όταν θα ξεσπάσει πίνα, μήπως μαζεύει από θέματα. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Για να δούμε Ακριβώ πω έχουν τα πράγματα που είναι αρκετά περιπλοκά όσον αφορά τα κίνητα, τα κτίρια στο Λουξεμβούργο, όπως γνωρίζετε. Το ζώμονε το ιστορικό κοινοκτήριο τον καταλήψαμε γιατί είχε πρόβλημα με τον αμίαντο. Οπότε και έτσι ε, στις 15 Εβδόμου του 2014 το αποφάσισε επίσημη Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατόπιν ε, της γνωμοδότηση. Τη ε, αρχή του προπολογισμού, Οπότε θα έπρεπε να βρούμε κάποιου άλλους ε, χώρους για συνεδριάσεις, για γραφεία κλπ. Επίσης ε, αποθηκευτικούς χώρους, το ώστε να μπορέσουν να μετακομίσουν οι εργαζόμενοι εκεί οι υπάλληλοι. Κάτι το οποίο ήταν μια εξαιρετικού χαρακτήρα κίνηση. Οπότε είχαμε αυτές τις αποθήκες, τους χώρους που αναφέρατε και οπότε είχαμε 7.000 τετραγωνικά μέτρα, αποθηκευτικού χώρου και αυτό θα πρέπει να βρούμε. Όμω ε, κάναμε ένα εξορθολογισμό και χρειαζόμαστε τώρα λίγο, πολύ λιγότερο χώρο και αυτό το οποίο τώρα θέλουμε είναι να βρούμε ε, τα μισά, 3.500 τετραγωνικά μέτρα. Βέβαια αυτό είναι παλαιό θέμα γιατί ήδη υπήρχε σχετική ενημέρωση από τον Μάρτιο του 15 από την αρχή του προϋπολογισμού και τον ε, Σεπτέμβριο. Αυτό δεν ήταν καινούριο αίτημα, αλλά λοιπόν θα συνεχιστεί η αναζήτηση του χώρου που ακριβώ είχε επισημάνθει. Και οριστικά μετακομίσαμε το Ζωμονέ ναι, τέλος του Μαΐου του 17 τα κλειδιά επιστράφησαν στους κυρίους του κτίριου και επομένω έκλεισε η τέσσερα κοντά ιστορία. Οπότε με τον εξορθολογισμό τώρα είχαμε χαρακτηρισμό ε, αυτών των 20.000 αντικειμένων ε, και επίσης μπορούσαμε να εξορθολογιστούμε και σε σχέση με όλα αυτά τα αντικείμενα και ε, οπότε ε, είχαμε επίσης κάποιο χώρο για, τα, για την επιδιόρθωση των επίπλων και όλα αυτά, όλα αυτά όπως και άλλα αντικείμενα δόθηκαν στους παρόγνους σχετικών υπηρεσιών. Επίσης, έχουμε και τα θέματα της κτύπωσης. Ε, και έχουμε το Ντρόσπαχ και στο κτίριο Ντρόσπαχ το 9% θα αφορά τους χώρους για εκτύπωση ξηρές ουσίες στο 7%, άλλοι χώροι για γενική αποθήκευση, ε, για διάφορα είδη εξοπλισμού και επίσης ε, μεγάλο τμήμα αυτών των χώρων αφορούν την πληροφορική και κάποια εργαστήρια τα οποία χρησιμοποιεί η Γενική Διεύθυνση Πληροφορικής της Κομισιόν έγινε έρευνα αγοράς και κατελικά είπαμε ότι η πιο λογική λύση είναι να νοικιάσουμε και άλλους χώρους στο κτίριο Ντρόσμπαχ. Είναι θέματα συνέργειας, πολύ σημαντικά που ε, ήδη είχε γίνει στο Λουξεμβούργο με την υπηρεσία των δημοσιεύσεων που όπως ξέρετε είναι πολύ σημαντική υπηρεσία ε, οπότε τώρα συνομιλούμε με την υπηρεσία εκείνη για να δούμε τι θα γίνει στο μέλλον ούτω ώστε να μπορέσουμε το Ζων Μονέ 2 όταν θα είναι έτοιμο να χρησιμοποιηθεί για τους χώρους της εκτύπωσης που να χρησιμοποιηθούν και από ε, τις υπηρεσίες δημοσίευσης και όλα αυτά βεβαίω θα είναι διοργανικά επίσης από πλευράς των συνεργειών σας επισημαίνω ότι εδώ και χρόνια έχουμε τέτοιου συνεργασίες ε, ιδίω όσον αφορά τη, τους παιδικούς σταθμούς αλλά έχουμε και τα θέματα της ασφάλειας και είπαμε να κάνουμε κάποιο είδος κέντρου ελέγχου για τα οχήματα το οποίο και αυτό να είναι διοργανικό. Αυτό σαν πρώτη απάντηση. Τέλος πάντων, εδώ είμαι και ό,τι θέλετε ρωτήστε με. Ευχαριστούμε δεν ξέρουμε πολύ καλά τα πράγματα στο Λουξεμβούργο. Ξέρω ότι εφόσον είναι στην ημερήσια διάταξη μπορούμε να μάθουμε λίγο περισσότερα πράγματα σχετικά με τα προβλήματα. Το 2014 ήδη ε, έπρεπε να έχουμε πάει στο καινούριο κτίριο και το 2017 ακόμα δεν είναι έτοιμο. Επίσης, ε, τι γίνεται με τα τρόφιμα, πώς αποδικεύονται. η κυρία Χολμάιερ, θα πρέπει να μας πει κάποια πράγματα. Ναι, να πω ότι χαίρομαι ιδιαίτερα που η υπηρεσία έχει αφιερώσει ενέργεια για καλύτερο συντονισμό των πραγμάτων και δημοσιοποίηση της κατάστασης. Υπάρχουν κάποια ε, όμως ε, πράγματα τα οποία θα έπρεπε λίγο να τα διαλευκάνουμε. Τι γίνεται ας πούμε με τους εκτυπωτές. Χρησιμοποιούνται οι εκτυπωτές ε, του Κοινοβουλίου και καταλαβαίνετε ότι αυτά έχουν και κάποιες νομικές συνέπειες. Ε, το θέμα της ε, συνέργειας και της βελτιστοποίησης είναι ένα θέμα. Νομίζω λοιπόν ότι αν δεν είναι μεγάλη και βαριή οι εκτύπωτες, γιατί δεν είναι και τα τελευταία μοντέλα, είναι μοντέλα τα οποία είναι κάπως παροχημένα. Ναι, μεν λειτουργούν, αλλά δεν είναι και στα σημερινά στάνταρ της εκτύπωσης ε, βασικά. Όταν λοιπόν ε, ε, τα δούμε όλα αυτά, ίσως θα πρέπει να δούμε κατά πόσο έχει κάποιο νόημα να τα κρατήσουμε ή να πάρουμε καινούρια. Για το κτίριο Ζαν Μονέ να πω ότι πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί φέτος η Κομισιόν είπε ότι θα πήγαιναν όλα σύμφωνα με το σχέδιο. Αυτό ήταν λάθος από ό,τι φαίνεται και τελικά μιλώντας με τον Επίτροπο του είπα ότι αυτό δημιουργεί τη πιστεία στο Κοινοβούλιο. Γιατί υπάρχουν αυτές οι καθυστερήσεις, θα υπάρχουν ε, ε, περαιτέρω ε, επιβαρύνσεις, υπάρχουν φυσικά αυξήσεις στο κόστος. Γιατί και όπως ξέρει και ήδη η Κομισιόν, σε ένα working document ε, να γράφεις τέτοια πράγματα δεν είναι καλό, δεν δημιουργεί εμπιστοσύνη. Επίσης, ε, θα ήθελα πραγματικά να ξεκινήσουμε να προσπαθούμε με μεγαλύτερη διαφάνεια να βλέπουμε όλα τα ζητήματα, ειδικά για τα οικονομικά που είναι ευαίσθητα. Ε, συνεχώς ε, πρέπει να συνεργαζόμαστε σε επίπεδο λογιστικής, γιατί αυτή η συνέργεια θα μας βοηθήσει να βελτιστοποιήσουμε τα αποτελέσματα, να είμαστε πιο γρήγοροι, πιο αποδοτικοί και να είμαστε και ε, σε θέση ε, να κάνουμε ε, τις καθημερινές δραστηριότητες γιατί όπως είναι τα πράγματα τώρα δεν μπορούμε να αποθηκεύσουμε ούτε καφέ, ούτε συμπυκνωμένο γάλα, ούτε νερό. Ε, δεν υπάρχουν χώροι και πρέπει όταν μας τα φέρνουν να είναι ακριβώς τη στιγμή που τα χρειαζόμαστε. Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε λίγο πιο ξεκάθαροι ε, ως προς την προσπάθειά μας να βελτιώσουμε τις δομές ε, και να προσαρμοστούμε στις ανάγκες. Merci. Ευχαριστώ. Όσον αφορά στα τρόφιμα, έχω ήδη απαντήσει. Νομίζω ότι υπάρχει ένα ελάχιστο στόκ που πρέπει να είναι στη διάθεσή μας. Ε, υπάρχει λοιπόν αυτό το κομμάτι το οποίο είναι το ελάχιστο. Όσον αφορά στις συνέργειες, φυσικά συμφωνούμε ότι πρέπει να υπάρχουν συνέργειες ε, με το σύνολο των θεσμικών οργάνων. Είναι κοινό μας συμφέρον αυτό. Και φυσικά υπήρξαν δυσκολίες ε, ως προς την πλήρη χρήση των εγκαταστάσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Όμως τώρα είμαστε στη φάση που αυτό το Γραφείο Δημοσιοποίησης που είναι το ο επικεφαλής, ε, ο επικεφαλής ας πούμε, ε, θα βοηθήσει να βρεούμε τις κατάλληλες συνέργειες για τις καθυστερήσεις σχετικά με το κτίριο Ζάμονε 2. Έχουμε λάβει στα τέλη του 16, αρχές 17, αιτήματα σχετικά με την ασφάλεια, τους μηχανισμούς ασφαλείας. Ήταν πολύ σημαντικά ε, τα αιτήματα αυτά. Έπρεπε να τα μελετήσει το αρχιτεκτονικό γραφείο που έχει αναλάβει το κτίριο. Δεν είναι και φυσικά η Κομισιόν υπεύθυνη, είναι η διοίκηση των κτηρίων του κράτους του Λουξεμβούργου που είναι υπεύθυνη και πρέπει να συνεργαστεί και με τους αρχιτέκτονες. Αυτά τα μέτρα ασφαλείας έπρεπε να εξεταστούν λεπτομερώς και οδήγησαν σε συγκεκριμένες ε, επεκτάσεις των προθεσμιών κατά έξι μήνες. Για το κόστος θα μπορέσουμε να απαντήσουμε στις αρχές του επόμενου έτους, γιατί στα τέλη αυτού του έτους θα έχουμε το αναλυτικό σχέδιο του design και θα έχουμε και την αποτίμηση την οικονομική για το κάθε στοιχείο. Θα τα έχουμε, τα είχαμε ε, τέλη του καλοκαιριού όλα αυτά τα στοιχεία και δεν μπορέσαμε να ενημερώσουμε την αρχή του προϋπολογισμού για τις συγκεκριμένες καθυστερήσεις. Επίσης υπήρχε και ένα θέμα σχετικά με το ε, σημείο όπου θα χτιστεί το κτίριο. Συνεχίζω κυρία Πρόεδρε. Η εξκαφή λοιπόν ήταν ένα θέμα. Τον ε, Φλεβάρη θα έχουμε τη δυνατότητα να δώσουμε πιο αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τα προβλήματα που προέκυψαν σε αυτό το project. Το κτίριο Jean Monnet 2 όταν ολοκληρωθεί θα έχει κάποια χαρακτηριστικά πιο διαθεσμικά θα έλεγα. Για παράδειγμα θα έχει μία βιβλιοθήκη, ένα κέντρο συνεδριάσεων που στο οποίο θα έχουν πρόσβαση όλα τα θεσμικά όργανα και άλλες εγκαταστάσεις. Άρα είμαστε πλήρως υπέρ αυτής της λογικής ε, των διαθεσμικών συνεργειών. Αυτά είχα να πω κυρία Πρόεδρε να μιλήσουμε... μιλήσουμε για τις καθυστερήσεις στο κτίριο Ζαν Μονέ. Από πότε τα γνωρίζετε αυτά, ε, πώς παρακολουθείτε το project και πώς φροντίζετε να μην υπάρχουν περαιτέρω καθυστερήσεις, γιατί προφανώς οι καθυστερήσεις αυτές έχουν συνέπειες για την μεταβατική αυτή περίοδο ή μήπω εξ αρχής ήταν προγραμματισμένα έτσι τα πράγματα ε, και εμείς απλά δεν το έχουμε καταλάβει. Η συνάδελφος Χολμάιερ Κοιτάξτε, δεν σχετίζονται απαραίτητα τα δύο θέματα αυτό, γιατί από τη μία έχουμε θέμα ιδιοκτησίας ε, άλλων κτηρίων και εδώ να σας πω ότι αυτό δεν ε, το είχαμε ορίσει. Βρήκαμε ένα άλλο ε, κτίριο το οποίο δεν το ελέγξαμε. Γιατί δεν πήγαμε όμως εκτός Λουξεμβούργου. Αυτή είναι η ερώτηση που έχω να κάνω εγώ. Εφόσον τα τελευταία δύο-τρία χρόνια οι εργαζόμενοι υπάλληλοι δούλευαν υπό άσχημες συνθήκες που δεν είναι αποδεκτές. Και τότε λοιπόν το Κοινοβούλιο είχε συμφωνήσει και με το κτίριο Ντρόσπαχ, γιατί σίγουρα οι υπάλληλοι δεν θέλαμε να μείνουν υπό τις δυσχερείς αυτές ε, συνθήκες να δουλεύουν. Δεν δεχτήκαμε καμία κριτική γι' αυτό. Η κριτική έχει να κάνει πιο πολύ με το θέμα των αποθηκών. Έρχεστε και μας λέτε λοιπόν ότι σήμερα, τη σήμερα ημέρα χρειάζεται να αποθηκεύουμε τέτοιες ποσότητες αποθεμάτων τροφίμων. Τι να σας πω, νομίζω ότι κανένας από τον τομέα της γαστρονομίας δεν συμφωνεί. Τι να σας πω, νομίζω ότι είναι για γέλια. Το 80 που ήμουνα ε, μαθήτρια ε, είχαμε και τέτοιες αποθήκες. Ε, δεν λειτουργούν ε, όμως τα πράγματα έτσι σήμερα. Η γαστρονομία λειτουργεί διαφορετικά. Δεν τα κάνουμε αυτά. Δεν κρατάμε τρόφιμα 3 έως 6 μήνες στη γαστρονομία. Άντε να το κάνουμε αυτό με τα καλά ισπανικά ζαμπόν. Όχι όμως για τα αλεύρια, για τα καθημερινά αυτά προϊόντα. Εντάξει, άλλοι λόγοι είναι αυτοί που καθορίζουν πόσο πρέπει να φυλάσσονται και να αποθηκεύεται ένα προϊόν για να αναπτυχθεί η γεύση τους. Ε, όχι όμως και στα λεύρια, ούτε στον καφέ. Στο κτίριο Ζαν Μονέ, λοιπόν, να πω ξεκάθαρα ότι από αυτά που μας λέτε οι πληροφορίες που μας δίνετε είναι λάθος, είναι ασφαλμένες. και τα θέματα ασφαλείας στο κτίριο Ζαν Μονέ ήταν τουλάχιστον ένα χρόνο παλιά. Δεν μπορούμε να πούμε λοιπόν ότι δεν το γνωρίζαμε και γι' αυτό δεν το είπαμε στο Κοινοβούλιο. Αυτό πραγματικά δεν στέκει και δεν θέλω να κορδευόμαστε. Να μας πείτε ότι κάνετε λάθος μάλιστα, ότι θέλετε να τα παραχωρήσετε και να τα παραδώσετε όλα σε τέλεια κατάσταση, ε, εντάξει. Αλλά το είπε το ξέρατε, ε όχι, είπε το δέχομαι. και ότι έπρεπε να γίνουν αλλαγές για την ασφάλεια, για την ασφάλεια η οποία προέκυψε προφανώς και μετά τις επιθέσεις στις Βρυξέλλες προέκυψαν νέες προδιαγραφές. Α, μπορεί να υπάρχουν σωστοί λόγοι και δικαιολογημένοι, δεν λέω, αλλά μη μας λέτε δικαιολογίες ότι δεν το ξέρετε τότε. Το ξέρετε, μια χαρά το ξέρετε. Μπορεί να μην γνωρίζετε επακριβώς την έκταση. Εντάξει, εκεί σύμφωνοι. Αλλά στην περίπτωση αυτή μπορούσατε να πείτε στο Κοινοβούλιο θα κοιτάξετε για τους ε, χυψηλόγους ε, προέκυψε νέο σχεδιασμό να υπάρξει μια προειδοποίηση και στη συνέχεια θα ακολουθούσαν τα συγκεκριμένα αριθμητικά στοιχεία. Μάλιστα εκεί. Μέχρι τα μέση του έτους μας ανημέρωναν και μας έλεγαν ε, ότι όλα πήγαιναν καλά και όλα προχωρούσαν καλά, αλλά δεν επιπρόκειται να ελεκτροφεί το έργο όταν αναμένονταν εσά. Παρακαλώ λοιπόν, μη μας δίνετε ψευδοδικαιολογίες. Γιατί άλλως δημιουργείται ένα κλίμα ε, έλλειψης εμπιστοσύνης και αυτό πραγματικά με δυσκολεύει. Και ως εισηγήτρια για το θέμα αυτό με απασχολεί ιδιαίτερα αυτό. Και 7% ε, ε, της επιφάνειας της έκτασης και 9% της έκτασης με κόστος 1,7 εκατομμύρια το χρόνο είναι μεγάλο ποσοστό. Είμαι γενικά θετικό άνθρωπο, αλλά κάπου εξαντλείται και η ευγένεια. Γιατί θεωρώ ότι πραγματικά δεν μα δίνετε σωστέ πληροφορίε. Παρακαλώ. Όσον αφορά το Ζαν Μονέ 2 και τα μέτρα ασφάλειας, όπως σας είπα, ήταν πολύ αναλυτικές οι μελέτες, γιατί ήταν πολύ ε, δύσκολα ζητήματα τεχνολογίας εχμής. Ας πούμε το θέμα του πάρκινγκ, η είσοδη για τους υπαλλήλους και τους επισκέπτες. Αυτά έπρεπε να τα εξετάσουν λεπτομερώς στο αρχιτεκτονικό γραφείο. Και επαναλαμβάνω, στο τέλος του καλοκαιριού μάθαμε για το εύρος των καθυστερήσεων. Και δεν ήμασταν λοιπόν 100% έτοιμοι να κάνουμε μια πλήρη έκθεση για αυτά τα νέα δεδομένα. Θα έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε στα τέλη του έτους μόλις ε, τα νούμερα τα οποία θα αντιστοιχούν στο κόστος ε, για αυτές τις μετατροπές. Ίσως δεν ε, μπορέσαμε επαρκώς να προβλέψουμε τη σημασία αυτών των καθυστερήσεων, όμως όπως και να έχει ε, έχουν να κάνουν και με τον τρόπο που εκτελούνται οι εργασίες σε ένα εργοτάξιο. Να θυμάστε λίγο και άλλα ε, project. Υπήρξε μεγάλος ανταγωνισμός, είχαμε πολλά κομμάτια στο project. Τώρα για τα για το στόκ των τροφίμων να πω στην κυρία Χολμάγερ να έρθει να δει από μόνη της ότι τελικά ε, πρόκειται για κάτι περιορισμένο συνολικά και θα ήταν και μεγάλη μας χαρά να δει αυτή την διαχείριση. Ε, τόσο περιορισμένο δεν είναι. 1.700 τετραγωνικά μέτρα χώροι ε, για αποθήκες και 1.800 τετραγωνικά μέτρα για γραφεία, 3.800 ε, πραγματικά ε, είναι το μισό. Καταλαβαίνετε ότι αυτοί που εργάζονται στην πληροφορική το θαυμάζουν αυτό. δεν καταλαβαίνω πώς είναι δυνατόν να έχουμε με αυτή την τιμή αυτό το μέγεθος εγκαταστάσεων. Και γι' αυτό ε, πάντοτε ρωτάμε γιατί τα χρειαζόμαστε. Κυρία Πρόεδρε, όπως σας είπα και πριν, περάσαμε από τα 7.000 στα 3.500 τετραγωνικά μέτρα σε επίπεδο αποθηκών. Συνολικά μειώσαμε την επιφάνεια κατά 72%. Και αν να προσθέσουμε όλες τις επιφάνειες, όλα τα τετραγωνικά, δηλαδή στόκ, ε, εκτυπωτές, γραφεία και πληροφορική, φτάνουμε συνολικά στα 14, από τα 14.000 τετραγωνικά στα 4.000. Τεράστια εξοικονόμηση για την πληροφορική. Σας είπα ότι οι αποθήκες είναι παρόμοιες με αυτές ε, των ε, εστιατορίων, της εστίασης. Έχουμε ένα εργαστήριο για τη διεύθυνση όπου μπορούν να ελέγξουν το νέο εξοπλισμό. Αυτό δεν μπορεί να γίνει σε χώρους γραφείων. Όσον αφορά τους χώρους, ε, για, για την εστίαση είναι 270 ε, τετραγωνικά, ενώ ήταν 4.500. Αν θέλετε όλα αυτά τα νούμερα μπορούμε να σας τα στείλουμε και γραπτός. Ναι, ναι, αυτή την ε, προσφορά θα τη δεχτώ με μεγάλη χαρά μου. Η κυρία Χολμάγερ. Να πω λίγο κάποια πράγματα ε, σχετικά με τις δικές σας προτάσεις, ε, σύγχρονες, ε, σύγχρονη διαχείριση στοιχείων εστίασης υπάρχουν. Αυτές οι μέθοδοι ε, τις βλέπω και σε καντίνες και σε εστιατόρια. Για μένα δεν υπάρχει νόημα να έχουμε αποθήκες για τον καθένα. Ίσως καλό είναι να υπάρχει μια κεντρική αποθήκη ε, ή ε, τέλος πάντων ακόμα και μεταφορά από το ένα εστιατόριο στο άλλο. Οι κεντρικές αποθήκες δεν είναι πλέον τόσο σημαντικές όσο ήταν στη δεκαετία του 60. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να δούμε Καταρχάς, κατά πόσο για έξι ε, εστιατόρια πρέπει να υπάρχουν κεντρικές αποθήκες στο Λουξεμβούργο, υπάρχουν σύγχρονα συστήματα διοικητικής μέρημνας που μπορούμε να τα αποφύγουμε αυτά. Και να σας πω επίσης ότι ε, ε, είναι πολύ σημαντικό να πηγαίνω στο Λουξεμβούργο για τη σημασία της στήρησης αποθεμάτων δεν είπαμε κάποια πράγματα, απλώς είπαμε να υπάρχει ένας εγγεγραμμένος στόχος, ε, γιατί γενικά είναι κάτι φυσιολογικό ή κάτι ε, εξαιρετικός ε, να υπάρχουν τέτοια μεγάλα, τέτοια μεγάλη χώρη αποθήκευση στην Κομισιόν. Είναι κάτι που γίνεται συνήθως ή μια φορά στο τόσο. Αυτό που θα δούμε να κάνουμε είναι να εξορθολογήσουμε, να περιορίσουμε τις σχετικές ε, εκτάσεις των χώρων. Και τώρα λέμε για 4 για 4.400 ε, υπαλλήλους και άλλους εργαζομένους. Πρόκειται λοιπόν ε, για ένα αρκετά σημαντικό νούμερο, οπότε έχουμε λιγότερο από ένα τετραγωνικό αποθηκευτικού χώρου αναεργαζόμενο. Οπότε βλέπετε όλα αυτά είναι σημαντικά σημαντική τάξη μεγέθου. Όλα αυτά τέλο πάντων να σα τα διαβιβάσουμε και να δείτε ακριβώς τι αναλογεί. Αυτό που με ανησυχεί είναι ότι δεν κάνετε την προσπάθεια να μας αποντήσετε αν είναι απαραίτητο, γιατί δίνουμε χρήματα γι' αυτό. Θα μπορούσαμε να τα έχουμε κάπου αλλού. Το ερώτημα είναι αν είναι πραγματικά απαραίτητες αυτές οι αποθήκες τροφίμων, αν υπάρχουν πλεονεκτήματα το ερώτημα της αναγκαιότητας ε, είναι ένα θέμα που θα ήθελα να μας απαντήσετε και γραπτός και θα χαρούμε εάν η Κομισιόν ε, μπορεί να μας πει ε, σε αυτή την απάντησή της και κατά πόσο θα μπορούσαμε να έχουμε μια καλύτερη διαχείριση. Η κυρία Κάντεμπαχ, ναι, κοιτάξτε, δεν σας είχα δει. Λέει η κυρία Κάτεμπάχαν. Ε, καταλαβαίνω την κυρία Χολμάγερ ε, με το θέμα της γαστρονομίας, όμως όλα αυτά έχουν να κάνουν λίγο και με την προστασία από τις καταστροφές, με την πρόληψη, ε, δηλαδή τσάι, ρύζι, γάλα είναι κλασικά πράγματα τα οποία έχουμε για τη διαχείριση καταστροφών. Και αυτή είναι η ερώτησή μου τώρα στην Κομισιόν. Αν πίσω από αυτό το θέμα της στήρησης αποθεμάτων έχει να υπάρχει αυτή η λογική της διαχείρισης καταστροφών. Ναι, παρακαλώ, για να δούμε λίγο το Λουξεμβούργο τι έχει να πει. Πολλές φορές έχουμε χιονοδιέρες, αλλά... Εκτός μικροφώνου. Εντάξει, χαιρόμαστε τώρα που για τους 4.000 εργαζόμενους υπάρχει τέτοια πρόβλεψη. Τι κάνουμε τώρα, περιμένουμε τις γραπτές πληροφορίες σας από την κυρία Χολμάγερ. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η εμπειρία να εξετάσουμε μαζί σας αυτή την έκθεση. Θα μπορούσατε γενικά να μας δώσετε και μια επισκόπηση των χώρων των γραφείων και ποιοι είναι ποιος είναι ο αριθμός ε, των υπαλλήλων που είναι εκεί και πόσο κοστίζει και το ενίκιο σε κάθε κτίριο αναέτος και ανατετραγωνικό. Όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά στοιχεία για τη δική μας δουλειά. Ευχαριστώ. Θέλετε να πείτε κάτι άλλο για να κλείσουμε. Απλώς ότι βεβαίως και υποσχόμαστε να σας δώσουμε όλες τις πληροφορίες που χρειάζονται και να είναι τα στοιχεία όσο είναι πιο ενδελεχή. Να θίξω ένα θέμα για άλλη μία φορά. Ε, σας ευχαριστώ Ευχαριστώ για τις ε, προσπάθειες που κάνατε να μας ενημερώσετε. Ήταν πολύ καλή η συνομιλία με τους ε, υπαλλήλους, όμως ε, θα πρέπει και στην Επιτροπή Προϋπολογισμού να γνωρίζουμε ποιες είναι οι αλλαγές για το κτίριο Ζανμονέ 2, όχι ως working paper, να δούμε αν μπορούμε να μείνουμε σε αυτό το 10% ή να πάμε πέρα από αυτό. Γιατί μέσα στο 10% δεν χρειάζεται να υπάρχει ενημέρωση, αλλά μετά το 10% ε, υπάρχουν, υπάρχει υποχρέωση ενημέρωσης. Υπάρχει αυτή η απόφαση και δεν πρέπει να την ξεχνάμε. Με χαρά μας ε, θα δεχτούμε οποιαδήποτε δουλειά γίνεται στην Επιτροπή Προϋπολογισμού για να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε τα στοιχεία για την απαλλαγή. Με αυτά φτάσαμε στο τέλος αυτού του σημείου της ημερήσιας διάταξης. Σας ευχαριστούμε πολύ. Πάμε τώρα στο σημείο 9. Είναι εδώ η συγκήτρια. ειδικη Ειδική έκθεση αριθμός 10-2017 του Ευρωπαϊκού Ελεκτικού Συνεδρίου Απαλλαγή 2016 στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, προς τους νέους γεωργούς η, η κυρία Κάντεμπαχ είναι η εισηγήτρια και έχει το λόγο. Uh, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, μου δώσατε την ευκαιρία να σας παρουσιάσω αυτή την έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου που έχει τον τίτλο Κοινοτική στήριξη σε νέους ε, γεωργούς. Θα πρέπει να είναι καλύτερα στοχευμένοι ούτως ώστε να υπάρχει πραγματική ανανέωση και διαδοχή των γενναιών επί τη βάση κάποιου γνώμη και uh, Και βλέπετε ότι έγινε αυτός ο έλεγχος η συνεργασία επιτροπής και κράτων μελών εκείνων που έχουν ε, την ε, ε, που είναι επιλέξιμα τέλο πάντων για τέτοια κονδύλια Γαλλία, Ιταλία, Πολωνία και Ιταλία. Πρόκειται για το 56% του συνόλου των πόρων που στοχεύουν εις τους νέους γεωργούς. Και τα ποσά αυτά είναι 10 δις σε διάστημα ε, ξεκινάμε από το 2007 μέχρι το 2013, δύο δημοσιακές προοπτικές δηλαδή, 3,2 δις ήταν τότε και αφορούσε τον πυλώνα υπαριθμών 2 και το 14 με 20 το αντιστοιχό ποσό το οποίο έχει καθοριστεί είναι 6,4 δις. 3,8 για τον δεύτερο πυλώνα και 2,6 για τον πρώτο πυλώνα. Για τον οικονομικό έλεγχο ασχοληθήκαμε με το ζήτημα του κατά πόσον η κοινωτική στήριξη είναι σωστή, ούτω ώστε να βοηθά αποτελεσματικά και να βελτιώνεται η κατάσταση όσον αφορά την ε, διαδοχή της μιας γενιάς από την άλλη. Αυτό, αυτό είναι το κλειδί στην υπόθεση αυτού του ελέγχου, γιατί αυτή η ανανέωση από πλευράς γενναίων είναι ο βασικός στόχος της στήριξης προς τους νέους γεωργούς. Και Μόλις ολοκληρωθεί ο οικονομικός έλεγχος θα δοθεί η απάντηση κατά πόσον έχουμε αυτή την ανανέωση. Δεν έχουν προφηθεί όλα, συνεχίζεται τέλο πάντων η εκταμείευση και 10 δις ευρώ έχουν αφηρηθεί σε αυτήν την πρωτοβουλία αλλά ακόμα δεν είδαμε, δεν παρατηρήθηκε ανανέωση πλευράς Έχουμε τώρα αυτή την ε, παρουσίαση, βλέπετε τις διαφάνειες, πολύ σημαντική ε, ε, εικόνα που βλέπετε τώρα, διότι δείχνει τα αποτελέσματα της στήριξης των νέων γεωργών στην περίοδο 2005 έως 2013. Η μπλε γραμμή δείχνει τον αριθμό των νέων γεωργών στην Ένωση. Μειώθηκε κατά αυτή την έννοια αιτία 5 με 13 από 3,3 εκατομμύρια έφτασαν στα 2,3 εκατομμύρια. Χάσαμε ένα εκατομμύριο νέους γεωργούς. Οπότε αυξήθηκε το πόσο γη κατέχουν οι Νέα Γεωργία από 19 εκτάρια ανέβηκε στα 24. Είναι η κόκκινη γραμμή. Άρα, λιγότερη γεωργή, μεγαλύτερες εκτάσεις. Πρόκειται για ευρύ για κατηγορία, γιατί πρόκειται για κάποιους γεωργούς οι οποίοι είναι κάτω των 45 ετών και συρρυκνώθηκε η έκταση που έχουν από 57,7 το 2005 έφτασε 57,9 το 2013. Πρόκειται για μια γενικότερη εικόνα του τοπίου και το πρόβλημα είναι γενικότερο δεν είναι μόνο θέμα νέων γεωργών αφορά γενικότερα την Ευρωπαϊκή Γεωργία ότι χάνονται, χάνουμε ε, εκμεταλλεύσεις. Βλέπετε, στην περίοδο 2007, σύγχρονα 2005 έως 2013 διορθώνει ο μιλητής, ο αριθμός των εκμεταλλεύσεων στην Ένωση μειώθηκε από 14,5 σε 10,7. Πάντα μιλούμε για εκατομμύρια εκμεταλλεύσεων. Άρα χάθηκαν σχεδόν 4 εκατομμύρια εκμεταλλεύσεις κατά την σχετική δεκαετία. Επομένως, 400 επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις τέλος πάντων, ανά έτος. 30.000 το μήνα, 10.000 την ημέρα. Ε, αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα και θα πρέπει να ληφθεί υπόψη στην συζήτηση που πρέπει να γίνει για την κοινή ερωτική πολιτική στο πόσο θα κρατήσει αυτή η πορεία, γιατί θα πρέπει να γίνει για να την φρενάρουμε. Άρα, αυτό αφορά και το σύνολο του αριθμού των εκμεταλλεύσεων που έχει συρρυκνωθεί και έχει συρρυκνωθεί, είπαμε, και ο αριθμός των ε, νέων γεωργών. Επόμενη διαφάνεια. Σε αυτή τη διαφάνεια μπορείτε να δείτε πόσο σοβαρό είναι το πρόβλημα. Είναι πρώτα πρώτα η γκρίζα γραμμή κάτω-κάτω που δείχνει το ποσοστό των νέων γεωργών σε σχέση με το συνολικό αριθμό γεωργών. Είναι 20 έως 21% είναι οι γεωργοί. Οι γεωργοί που είναι κάτω των 45 όπως είπαμε. Και είναι το ίδιο το ποσοστό των νέων σε σχέση με το σύνολο των εργαζομένων. Περίπου 50% των εργαζομένων. Και ε, λέμε και είναι η πράσινη γραμμή στην κοινωνία πώς είναι οι εργαζόμενοι και πώς είναι οι νέοι των 45% 45% λοιπόν γενικώ και 20-21% όσον αφορά τους νέους γεωργούς και τη γεωργία. Και κατά αυτή την ε, περίοδο 2007-2013 η συμμετοχή των νέων γεωργών σε σχέση με το σύνολο των γεωργών έπεσε από 21,8% σε 21,3%. Επομένω, δεν υπήρξε εδώ πέρα ανανέωση γενναιών, η κατάσταση επιδεινώνεται σε σχέση με προηγουμένω. Δεν ξέρω πόσο ευκρινής είναι αυτή η εικόνα αυτός ο πίνακας, αν να σας τα εξηγήσω. Πρόκειται για την ε, διάρθρωση του θέματος ε, των γεωργών στα κρατημέλη. Μπορείτε να παρατηρήσετε κάποιες μικρές βελτιώσεις βελτιώσεις. όμως μόνο συγκεκριμένα κρατημέλη. Βουλγαρία, Εστονία, Ιταλία, Σλοβενία, Σλοβακία. Πολωνία. αυτά. Κατά τα λοιπά. Μπορεί να παρατηρήσει κανείς. Επιδείνωση της κατάστασης σχέση με Για παράδειγμα, στη Γαλλία. Το ποσό των νέων γεωργών σχέση με το σύνολο των γεωργών συρρυκνώθηκε από 32% στο 28% στην Γερμανία. Αλλά η Γερμανία ε, δεν είχε στήριξη στην περίοδο 7 έως 13 μόλις 2 εκατομμύρια ευρώ εκταμιεύτηκαν αλλά και εκεί μειώθηκε το ποσοστό των νέων γεωργών από το 36% κατέβηκαν στο 26% του συνόλου των γεωργών. Αυτό σημαίνει πολύ σοβαρό πρόβλημα ε, όσον αφορά το ηλικιακό των γεωργών. Επίσης σε αυτόν τον πίνακα μπορείτε να διαπιστώσετε ότι οι πιο νέοι γεωργοί κάτω των 35 ε, μόνο σε δύο κράτη-μέλη αυτή η κατηγορία κάτω των 35 είναι άνω του 10% στην Αυστρία και στην Πολωνία δεξιά βλέπετε τι γίνεται με τους πιο ηλικιωμένους από τους Γιώργους. Αυτούς λοιπόν είναι άνω των 65. Μόνο σε τρία κρατημέλη αυτή η κατηγορία είναι κάτω του 10% Γερμανία, Αυστρία και Πολωνία. πάνω των 40% στην Πορτογαλία είναι πάνω του 50%. Άρα οι περισσότεροι γεωργοί στην Πολωνία είναι άνω των 65%. Βέβαια διαφέρει ανακράτωση η κατάσταση. Αυτό σημαίνει ότι ο καθένας έχει άλλο πρόβλημα όσον αφορά το ηλικιακό των γεωργών. Υπάρχουν κάποια κοινά προβλήματα όλη την Ευρώπη, αλλά γενικό μπορούμε να πούμε για το συγκεκριμένο θέμα διαφέρει η κατάσταση ανά χώρα. Άρα άλλη λύση χρειάζεται η κάθε χώρα. Θα πρέπει να επιδείξουμε ευελιξία μια που η κατάσταση διαφέρει από χώρα σε χώρα. Εδώ βλέπετε πόσο απορροφούνται οι πόροι ε, Οικονομικός έλεγχος έγινε στους τέσσερις του χρήστες, <coughs> Γαλλία, Ιταλία, Πολωνία, μεταξύ αυτών και τώρα. Μάθετε τη λογική της παρέμβασης. Πολύ σημαντικό το ότι δεν βρέθηκαν ε, καταχρήσεις, ε, παρατυπίες όσον αφορά τους επιλέξιμους γεωργούς. Μα είναι η λογική της ε, παρέμβασης και μπορείτε να δείτε τη σελίδα 34 στην έκθεσή μας και εκεί έχουμε παραθέσει κάποια παραδείγματα. Φερρυπίν, η ενίσχυση για τους γεωργούς που έχουν 500 εκτάρια. Αυτοί δικαιούνται 100.000 ευρώ ως ε, άμεση πληρωμή και επιπλέον 3.000 ε, εάν πρόκειται περί νέου Γιώργου. Να, η, ε, ενίσχυση. Όμως δεν υπήρξε κάποιο είδου επίπτωση για την ανανέωση των γενναιών. Επίσης, βοηθήσαμε κάποιους που ήταν εταίροι ε, και είχαν ας πούμε συμμετοχή στην σχετική εταιρεία 16%. Δεν ήταν ενεργοί γεωργοί, αλλά και αυτοί έλαβαν ενίσχυση ύψους 4.000 ευρώ. Ούτε σε αυτό το μέτωπο είχαμε κάποιο είδου θετικές επιπτώσεις για την των γενιών. Τέλος, οι συστάσεις μας. επόμενη διαφάνεια. Μισό λεπτό να βρούμε τη σωστή διαφάνεια. Όχι, θα κάνουμε εδώ πέρα παρουσίαση ε, του ελέγχου και των λεπτομεριών, αλλά οι, ποιες είναι οι προτάσεις. Πρώτα πρώτα να βελτιωθεί η λογική της παρέμβασης και να ενισχύσουμε την αξιολόγηση των αναγκών. Δεύτερον, να βελτιώσουμε τη στόχευση των μέτρων και η τρίτη σύστασή μας είναι να βελτιώσουμε την εποπτεία, τον έλεγχο και την αξιολόγηση. Επίσης να ευχαριστήσουμε την κυρία Κάντεμπαχ για το κείμενό της. Ευχαριστούμε που συνέβαλε στι συστάσει μα. Πολύ σημαντικό αυτό για τι συζητήσει που θα γίνουν στο μέλλον. Οι συζητήσει για το μέλλον τη κοινή αγροτική πολιτική όσον αφορά το χρονικό διάστημα μετά το 2020. Πολύ σημαντικό να καθορίσουμε ποια θα είναι η λογική των ε, επεμβάσεων για μια πραγματική ανανέωση των γενιών. Γιατί τώρα τα χρήματά μας δεν πιάνουν τόπο. Δεν υπάρχει ανανέωση γενιών. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και πραγματικά η έκθεση είναι πραγματικά πάρα πολύ καλή ποιότητα και είναι και σημαντική η έκθεση. Γι' αυτό λοιπόν και μπήκε στην ημερήσια ε, διάταξη δεδομένων και των προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε. Θα πρέπει να συζητήσουμε λοιπόν τι θα κάνουμε. Το λόγο έχει η συγκεκριμένη Κυρία παρακαλώ. Σα ευχαριστώ. Και να ήθελα να συγχαρώ και να ευχαριστήσω τον συνάδελφο, τον πρώην συνάδελφο, ε, ε, για την δουλειά του και να δώσω κάποια αριθμητικά στοιχεία για να καταδείξω πόσο έντονη είναι η κατάσταση και πόσο δραματική είναι η κατάσταση σε ό,τι αφορά και τις συστάσεις τις οποίες θα προβούμε. Καταρχάς, ο αριθμός των νερών έχουν ε, μειωθεί από τρία 2,3 εκατομμύρια σε 2,2 το 2005 στο 2013. Επίσης, ε, παρά το γεγονός ότι οι χερσαίες εκτάσεις παρέμειναν οι ίδιες, μειώθηκε ο ρυθμός των γεωργών. Και αυτό φαίνεται και από την έκθεση. Εξετάζοντα πιο λεπτομερό τα στοιχεία αυτά, διαπιστώνουμε ότι οι καταστάσεις είναι πάρα πολύ διαφορετικές από κράτος μέλος σε μέλος και Μάλιστα και από περιφέρεια. Σε περιφέρεια υπάρχουν πολλές ιδιαιτερότητες. Γενικά εγώ είμαι υπέρ, γιατί πιστεύω ότι είναι και πιο απλό για, την, ε, τον έλεγχο. Αν θέλουμε λοιπόν να πετύχουμε το στόχο της ανανέωσης των γενιών, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε μέτρα στην προκειμένη περίπτωση θα αντιμετωπίζουν τα συγκεκριμένα προβλήματα που έχει κάθε περιφέρεια. Το σχέδιο της χρηματοδοτήσης ε. Το κοιτάξτε και οι συνάδελφοι. Θα ήθελα να συμφωνήσω και με τι συστάσει ε, του Ελληνικού Συνεδρίου. Τέσσερι ε, προσθήκε στα εφιστάμενα μέτρα ε, στα πλαίσια τη ΚΑΠΑ. Καταρχά, όλα τα μέτρα τα οποία χρησιμοποιούνται για την υποστήριξη θα πρέπει να αξιολογηθούν σε βάθος. Αυτό προέκυψε νομίζω από τη σύγκριση ότι από τη μία θέλουμε μια συγκρισιμότητα σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και το γεγονός ότι κατά πόσον οι δείκτες αυτή απόδοση είναι συνεκτική ομογενής ή όχι, είναι σημαντικό. Δεύτερη σύσταση. Εμπόδια, προσκόμματα. Τι προσκόμματα αντιμετωπίζουν τα κράτη-μέλη. Τι εμποδίζει τους νέους από τον να προχωράνε τις επιχειρήσεις. Και το θέμα των ε, συντάξεων. Και αυτό έχει σημασία για την ανάληψη των επιχειρήσεων. Η πολιτική με το 2020 τώρα. Πώς θα πρέπει να δημορφωθούν τα πράγματα. Υπάρχουν πολιτικά μέσα τα οποία μας τα επεξήγησε και ο συναδελφός και νομίζω ότι θα πρέπει να λεφθούν υπόψη διάφορα στοιχεία το θέμα των εμποδίων όπως είπαμε αλλά και το θέμα των συγκεκριμένων αναγκών το θέμα των νεοφυών επιχειρήσεων και των ε, νέων επιχειρηματιών κατά πόσον πρόκειται για πολιτικά ζητήματα, κατά πόσον πρόκειται για συγκεκριμένα ζητήματα γεωργικά. Και με τι πολιτικά μέσα μπορούμε να προωθήσουμε την ανάληψη επιχειρήσεων. Τι χρειαζόμαστε λοιπόν στα διάφορα κράτη-μέλη για να τι πιο εύκολη η ανάληψη και παράδοση επιχειρήσεων. Βλέπουμε ότι υπάρχουν ε, ένα ποσό ε, κατά ε, ενισχύσεων που θα πρέπει να καταβληθούν, θα πρέπει να είναι στόχοθετημένα. Ποιο μέτρο λοιπόν, ποιο μέτρο υποστηρίξης, ποιο οικονομικό μέσο ανταποκρίνεται καλύτερα στην εκάστοτε ανάγκη. Ένα άλλο σημείο το οποίο προκύπτει από την έκθεση. Χρειαζόμαστε πιο πολλές πληροφορίες, ε. θέματα δηλαδή, πληροφορίες για την ε, ενδεχόμενη υποστήριξη, ενδεχόμενες μορφές υποστήριξης σε ό,τι αφορά και τους, ε, τη διαδοχή των επιχειρήσεων, μέσα τα οποία μπορούν να τα συνεχίσουν, να συνεχίσουν να ωφελούνται και οι νέοι επιχειρηματίες και οι νέοι γεωργοί σε ό,τι αφορά τώρα τα μέτρα, πώς προσανατολίζονται τα μέτρα σε κάθε κράτος μέλος. Σαφή κριτήρια, γιατί διαπιστώσαμε στην έκθεση ότι τα κριτήρια προφανώς ερμηνεύονται με διαφορετικό τρόπο κατά περιοχή. Και τέθησε και συγκεκριμένο το ερώτημα, πώς μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι οι ενισχύσεις πραγματικά έχουν σκοπό τον νερό γεωργό, ο οποίος ασχολείται α, κατά κύριο λόγο με την αγροτική εκμετάλλευση. Θέλουμε λοιπόν καλύτερα ελάχιστα πρόγρα, πρότυπα, ελάχιστες προδιαγραφές. Και άλλο ένα πρόβλημα το οποίο προκύπτει είναι το θέμα της κατάλληλης συμπληρωματικότητας των μέσων. Δηλαδή, να μην εξαντλούνται, αν θέλετε, τα μέσα τα πρώτα χρόνια και να μην διατίθεται τελικά τίποτα τα τελευταία χρόνια της προγραμματικής περίοδου. Τέταρτο σημείο το οποίο θέλω να θίξω. Οι ομοθετικέ προδιαγραφέ για την περίοδο μετά το 2020 σε ό,τι αφορά το συνολικό σύστημα έλεγχου και επιτήρησης. Αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο παρουσιάζεται σε σχέση με τις ενισχύσεις στον αγροτικό τομέα και στα διαφορετικά ταμεία, ότι ουσιαστικά δεν υπάρχουν συγκρίσιμα στοιχεία και κάτι γενικό για το περιεχόμενο της έκθεσης. Και μας απασχολεί ιδιαίτερως. προβληματικό στοιχείο το οποίο σχετίζεται με το θέμα αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με το οικονομικό σκέλος και το πολιτικό σκέλος της αγροτικής πολιτικής. Πρόκειται για ένα ζήτημα το οποίο το αντιμετωπίζουμε από κοινού με άλλους κλάδους σε ό,τι αφορά την ύπεθρο, σε ό,τι αφορά τις περιοχές όπου λαμβάνει χώρα η αγροτική εκμετάλλευση, αλλά θα πρέπει αυτό να αποτελεί, ξέρετε, και ένα χώρο βιώσιμο για όσους εργάζονται εκεί. Χρειάζεται κοινωνική ασφάλιση, χρειάζεται επίσης ε, προβλέψεις για τους ε, ε, συντρόφους των ατόμων αυτών που δεν ασχολούνται με τη γεωργική εκμετάλλευση και ενδεχομένως θέλουν να ασχοληθούν και ζουν στην Ήπεθρο. Πρέπει η ζωή λοιπόν στην Ήπεθρο να διαμορφωθεί με πιο ελκυστικό τρόπο. Αυτό θεωρώ ότι θα βελτιώσει σημαντικά την κατάσταση. Δεν αρκούν δηλαδή και μόνο τα οικονομικά κίνητρα όπως διαμορφώνονται σήμερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να ορίσουμε και τον κύριο Σικέρσκι, τον ε, πρόεδρο της Επιτροπής Γεωργίας. Και άλλους συναδελφούς είχαμε καλέσει από την Επιτροπή Γεωργίας. Νομίζω ότι είναι λάθος αυτό που μας είπε το ελεκτικό συνέδριο. Το κοινοβούλιο μετά γιατί έβαλε ως ανταμοιβή, αν θέλετε, 34 εκατομμύρια για την επόμενη περίοδο. Τι θα κάνουμε λοιπόν για να τα βάλουμε όλα αυτά στη σειρά και να φροντίσουμε πραγματικά να υπάρξει αλλαγή των γενεών στη Γεωργία. Αυτός είναι ο στόχος μας. Γιατί στην παρούσα φάση ε, τα μέσα έχουν ε, λειτουργήσει μόνο σε επιδοτήσεις. Και αν δεν αλλάξουμε κάτι, εκεί θα μείνουν, σε αυτό το επίπεδο. Δεν υπάρχει κάποιος ε, ενεργός προσανατολισμός. Και θεωρώ ότι αν συνεχίσουμε έτσι, ουσιαστικά χάνει το κύρος της όλες οι επιδοτήσεις και οι ενισχύσεις. Η κυρία Σμιτ. Ναι, ευχαριστώ τη συνάδελφο Κάντεμπαχ. Αυτά που είπατε κι εσείς κυρία Πρόεδρε και η συνάδελφος είναι πράγματα στα οποία θα ήθελα να προσθέσω κι εγώ κάτι. Η ανάλυση των αναγκών είναι η λέξη κλειδί δεν μιλάμε μόνο για το που υπάρχουν νέοι, αλλά και για το που στέλνουμε τα χρήματα και τελικά εάν ε, τα χρήματα πηγαίνουν εκεί που ανήκουν ή τελικά κάποιοι νέοι παίρνουν δύο φορές και τρεις φορές χρήματα και άλλοι καθόλου. το εισόδημα των νέων γεωργών, πόσο αποδοτικές είναι οι επιχειρήσεις τους, ποια είναι τα ποσοστά, οι για την ε, εναλλαγή των γενεών. Υπάρχουν συγκεκριμένα ερωτήματα προς την Κομισιόν. Είναι δικαιολογημένο που δεν υπάρχει η ανάλυση των αναγκών για το που δίνονται τα κονδύλια. Επίσης, για παράδειγμα, πώς μπορούν τα χρήματα από τον πρώτο πυλώνα για την εναλλαγή των γενεών να ε, δοθούν σε κάποιον ο οποίος έχει μία γεωργική εκμετάλλευση. Επίσης, τα κράτη-μέλη θα πρέπει να έχουν μια γενικότερη εικόνα για το ποια είναι τα κονδύλια ε, τα οποία εξασφαλίζονται σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Ε, πριν μπορεί κανείς να δράσει πρέπει να κάνει ανάλυση. Επίσης, ποια είναι τα κριτήρια επιλογής ε, και πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν καλύτερα στο δεύτερο πυλώνα, έτσι ώστε να ενισχύσουμε τα καλύτερα project. Για... Οι πληροφορίες σε αυτό το επίπεδο είναι πάρα πολύ σημαντικές. Δεν μπορούμε οι επιδοτήσεις να δίνονται στην αρχή και μετά να μην υπάρχει τίποτα. Υπάρχει λοιπόν δυνα... Ε, ανάγκη να δράσουμε. Υπάρχουν πάρα πολλές πληροφορίες που μας δίνονται μένα, αλλά πρέπει να είμαστε πολύ συγκεκριμένοι και να έχουμε μια πρόταση για βελτίωση στα χέρια μας. Ε, ζητώ λοιπόν από την Κομισιόν να υποστηρίξει το ελεγκτικό συνέδριο και να μας δώσει πληροφορίες ε, οι οποίες ακριβώς ε, θα λένε που πρέπει να πηγαίνουν τα χρήματα. Επόμενος, ο συνάδελφος Ζαμπάμα. Ευχαριστώ πολύ, ειδικότερα τον κύριο Μακεκόφσκι από το ελεγκτικό συνέδριο που μας παρουσίασε μια πολύ καλά δομημένη και ξεκάθαρη έκθεση. Υπάρχουν συγκεκριμένες ε, παρατηρήσεις και απτές συστάσεις στην έκθεση. Και φυσικά να ευχαριστήσω και την εισηγήτρια την κυρία Κάντανμπαχ. Συμφωνώ σχεδόν με όλα όσα είπατε. συζητούμε συγκεκριμένα τους νέους γεωργούς εδώ, που είναι πολύ σημαντικό, διότι όπως βλέπετε, σε κάποιες από τις μεγαλύτερες αγροτικές χώρες ο πληθυσμός των γεωργών γυράσκει ταχαίως. Και δεν είναι και πολλοί νέοι που θέλουν να διαδεχθούν σε αυτή την πολύ δύσκολη σκληρή δουλειά. Παρά τα εκατομμύρια και τα δισεκατομμύρια που τους δίνουμε, η ίδια η δουλειά δεν ανταποδίδει. Όσον αφορά τώρα στις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης όμως, να πω ότι ήταν καλές για δεκαετίες, αλλά το 2017 πλέον ε, ε, είναι απίστευτο να έχουμε ένα σύστημα και μιλάω συγκεκριμένα για τον πρώτο πυλώνα το οποίο από την έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου φαίνεται πως απλώς δεν έχει πλέον νόημα. Δεν υπάρχει γενικότερη αξιολόγηση των αναγκών. Αυτό έχει να κάνει με τους νέους γεωργούς, αλλά το θέμα πάει παραπέρα, πάει γενικότερα στον πρώτο πυλώνα είναι υπερτυποποιημένο, ε, οι στόχοι ε, δεν ε, αντικατοπτρίζουν τη γενική στόχευση για ανανέωση των γενεών, εναλλαγή των γενεών. Γενικά υπάρχει ανάγκη για δραματική αναδιάρθρωση του πρώτου πυλώνα. Έχω εξετάσει το θέμα προσεκτικά εδώ και πολύ καιρό. και εξετάζοντας και την κατάσταση με το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο μετά το Brexit, πραγματικά βλέπουμε ότι υπάρχει ανάγκη για δραματική ε, αλλαγή της κατάστασης. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να περικόψουμε την ΚΑΠ, αλλά τα χρήματα που δίνονται πρέπει να δίνονται πιο υπεύθυνα και πρέπει να αποδεικνύουμε και τα αποτελέσματα. Αν δεν βλέπουμε αποτελέσματα από τις επιδοτήσεις ε, στους γεωργούς οι οποίοι παίρνουν εκατομμύρια το χρόνο, κάτι πρέπει να κάνουμε, να αναδιοχετεύσουμε τα χρήματα. Και αν κατάλαβα καλά από τα προκαταρκτικά στοιχεία που μας έδωσε η Κομισιόν, ε, θα είναι πολύ ενδιαφέρον το μέλλον. Ε, θα ήθελα να ρωτήσω την Κομισιόν εάν βλέπουν την ανάγκη να υπάρξει πραγματικά μια δραστική αλλαγή στον τρόπο που αλληλεπιδρούν ο πρώτος και δεύτερος πυλώνας στα κράτη-μέλη. Πώς θα μπορέσουμε να δώσουμε στα κράτη-μέλη μεγαλύτερο λόγο στον τρόπο χρήσης και αποδοτικής και αποτελεσματικής χρήσης των χρημάτων. Ενώ ταυτόχρονα βέβαια θα έχουμε και πιο ισχυρά κριτήρια για, το, για τα αποτελέσματα. Πρέπει τα αποτελέσματα να φαίνονται. Πολλές φορές και εκ των προτέρων. Μιλάμε συνεχώς για τα ίδια πράγματα. Γυρίζουμε γύρω από τα ίδια πράγματα όταν μιλάμε για τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά όταν ε, μιλάμε για αυτά τα θέματα, πολλά ζητήματα πρέπει να εξετάζουμε ταυτόχρονα και όχι ένα μόνο θέμα. Ένα από τα προβλήματα που έχουμε στον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό είναι ότι τίνουμε να επικεντρωνόμαστε σε κάθε πράγμα ξεχωριστά κάθε φορά και δεν βλέπουμε τη γενικότερη εικόνα επαρκώς τουλάχιστον. Όσον αφορά λοιπόν στους νέους γεωργούς, ναι, είναι πολύ σημαντικό, αλλά δεν μπορεί να επιληθεί το θέμα αν δεν έχουμε στο μυαλά μας και την γενικότερη εικόνα της ΚΑΠ μετά το 2020 ε, αν δεν δούμε πώς θα χρησιμοποιηθεί ο πρώτος πυλώνας, πώς θα ζητούμε τα αποτελέσματα και πώς θα δαπανώνται ε, πιο καλά, ε, με πιο σόφρονα τρόπο τα χρήματα. Ευχαριστώ, συνάλφο Σίκιας και έχει το λόγο. Νομίζω ότι όλοι μας αναρωτιόμαστε τα ίδια πράγματα. Τα ίδια μας ερώτηση αναρωτήθηκε και η κυρία Κάντεμπαχ, αλλά και οι υπόλοιποι. Γιατί υπάρχει αυτό, ε, ποιος, ε, ποιο είναι το σκεπτικό γιατί ε, θέλουμε τα συγκεκριμένα αποτελέσματα και τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιώσουμε την κατάσταση περαιτέρω. Ξέρουμε ότι υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες προτιμήσεις σε κάποιες από αυτές τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις ε, και εταιρείε υπάρχουν ε, κάποιες σχέσεις μεταξύ των μελών των, της κάθε εταιρεία. Όμως αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε τελικά είναι να ξεπεράσουμε προβλήματα, γιατί υπάρχει έλλειψη ε, ε, εκτάσεων και επενδύσεων και η γη δεν πηγαίνει πάντοτε απαραίτητα στους γεωργούς. Αυτό είναι ένα γενικότερο πρόβλημα. Ήδη έχει υπάρξει μια σχετική έκθεση για τη συγκέντρωση γης στα χέρια λίγων. Πολλές φορές υπάρχει έλλειψη αρρώσιμης γης. Το ερώτημα λοιπόν είναι προφανώς το εισόδημα, τα έσοδα, έσοδα από γεωργικές επιχειρήσεις κατά 50% και 50% από άλλες δραστηριότητες και φυσικά τα ευρωπαϊκά κονδύλια και χρήματα. Ένα άλλο επίπεδο του προβλήματος έχει να κάνει με την ποιότητα διαβίωσης και το και των υποδομών στις γεωργικές περιοχές. Σε κάποιες περιοχές οι υποδομές ε, είναι πιο κακές. Σε άλλα κράτη-μέλη όμως δεν είναι και τόσο μεγάλο το πρόβλημα και όταν έχουμε νέους ειδικά που αναλαμβάνουν την επιχείρηση. Επίσης υπάρχει το ζήτημα των εργασιακών ευκαιριών σε αυτές τις περιοχές. Γιατί πραγματικά πρέπει να υπάρχουν και άλλες ευκαιρίες για εργασία. Ίσως πρέπει να είναι λίγο πιο πολύ εθνική η ε, αιρεσιμότητα, γιατί πολλές φορές έχουμε συγκέντρωση της γης. Πρόβλημα που έχουν πολλές χώρες και θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Αν δείτε λίγο το ευρωπαϊκό μοντέλο γεωργίας, το ερώτημα εδώ δεν είναι κατά πόσο θα πρέπει να μπορεί να επιβιώνει ο ισχυρότερος, γιατί όπως είπα υπάρχει η συγκέντρωση της γης και πρέπει να διασφαλίσουμε ότι οι γεωργοί έχουν κάποιο εισόδημα. Όλα αυτά πρέπει να τα έχουμε στο μυαλό μας. Ο παρακαλώ, Ευχαριστώ πολύ. Και ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η παρουσίαση. Πάρα πολύ σημαντικές πληροφορίες αυτές σε ό,τι αφορά την ε, καθορισμό της πολιτικής και νομίζω ότι ενώ ξοδεύουμε πολλά χρήματα δεν βλέπουμε να ανανεώνονται οι γενιές και αυτό που μας ανησυχεί ακόμα πιο πολύ στο πλαίσιο αυτό είναι το πώς θα δαπανηθεί τα υπόρρυγη σε ό,τι αφορά και τον Brexit, σε ό,τι αφορά α, τις πιέσεις που δεχόμαστε και οι τέτοιες εκθέσεις πρέπει να πω ότι είναι εξαιρετικές και δεν θέλουμε προφανώς να τιμωρήσουμε τον φόρο. Μας ανησυχούν ωστόσο ιδιαίτερα γιατί δημιουργούνται επιχειρήματα να σταματήσουμε να ξοδεύουμε λεφτά στην, στο πλαίσιο αυτό. Θα πρέπει λοιπόν κάπως να τα μαζέψουμε. Εγώ προσωπικά βρίσκομαι να συμφωνώ με το ΕΛΚ το που το λένε μεν εδώ αλλά όχι στις πατρίδες τους ότι τα χρήματα αυτά δεν κατανέμονται σωστά ουσιαστικά πηγαίνουν ε, στη βασίλισσα της Αγγλίας και όλα αυτά δεν είναι δικαιολογημένα προφανώς. Ε, κοιτάξτε, μπορούμε να τα περιπλέξουμε τα πράγματα ή μπορούμε και να τα απλοποιήσουμε. Ας πούμε ότι είσαι μαραγκός. Ως ε, οποιαδήποτε και να κλάβε και να είσαι όταν ξέρεις ε, δεν ε, πρόκειται να βγάλεις χρήματα. Πολύ απλά δεν πρόκειται να ξεκινήσεις το επάγγελμα αυτό. Τελικά ο κόσμος αυτό που θέλει είναι να βγάλει χρήματα, να μπορεί να ζήσει αξιοπρεπώς. Η Ευρωπαϊκή Ένωση προφανώ μπορεί να δώσει οικονομική υποστήριξη, αλλά θα πρέπει να υπάρχει και δεσποτική υποστήριξη. Νόμοθεσία που θα αποτρέψει τους μεγάλους ομίλους να βγάλουν χρήματα και από τη μήγα ξύγκη και τελικά να μείνουν οι χαμηλόμιστοι, αυτοί που είναι στο κάτω-κάτω μέρος της αλυσίδας, να μην έχουν τίποτα. και προφανώς όλοι θα πρέπει να προχωρήσουν προς τα μπροστά, αλλά και οι πιο ηλικιωμένοι δεν μπορούν να προχωρήσουν. Έχει γίνει λοιπόν μια αλλαγή από τότε που καταρτίστηκε η έκθεση και όπως θα μας πει και ο α, πρόεδρος της Επιτροπής Γεωργίας, εργαζόμαστε και για το πακέτο Omnibus και περιλαμβάνονται στοιχεία, ιδιαίτερα για τους νεαρούς ε, γεωργούς και για τις νεαρές οικογένειες. Υπάρχουν προβλέψεις. Αναρωτιέμαι όμω ποια είναι η απόψη τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. και του είσαι για το γεγονό ότι αφιερώσαμε κάτι στου νεαρού γεωργούς προκειμένου να έχουν δικαίωμα στα πέντε χρόνια το τόπο ακόμα. Αυτό είναι καλό, καλή είδηση. Αλλά μια χώρα όπως η Ιρλανδία, για παράδειγμα, βρίσκεται σε μια κατάσταση όπου δεν μπορούν να λαμβάνουν και τα πέντε χρόνια το ΠΑΠ. Αυτό πώς θα βοηθήσει τον οποιονδήποτε. Καταλαβαίνω ποια είναι η άποψη του Ελεκτικού Συνεδρίου και, για, και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι εφόσον δεν λειτουργεί καλά το σύστημα, πώς γίνεται. Μάλλον εφόσον λειτουργεί καλά το σύστημα, Πώ υπάρχουν χώρε μεταξύ των οποίων και η δική μου προ μεγάλη μου ντροπή που προσπαθούν να τα κλατώσουν και να μην δώσουν τα χρήματα αυτά. Καλή είναι η δουλειά και πραγματικά δεν θέλω να τιμωρήσω τον αγγελιοφόρο, αλλά όταν το μήνυμα τελικά περάσει προ τον έξω κόσμο δεν θα είναι θετικά τα αποτελέσματα. δεν θα κρυθούμε θετικά σε ό,τι αφορά θα δαπάνη των πόρων αυτών. Ευχαριστώ κύριε Σαλεμφράγκα. Σας ευχαριστώ πρόεδρε. Ευχαριστούμε και το Ελληνικό Συνέδριο για την έκθεση, ευχαριστούμε ε, και για το έγγραφο. Νομίζω ότι σε αυτή την έκθεση περιέχεται μια πολύ ενδιαφέρουσα ανάλυση για το τι γίνεται σήμερα με την κοινή αγροτική πολιτική στην ε, ε, Ένωση και για το συγκεκριμένο θέμα, δηλαδή την ανανέωση των γενιών και από ό,τι αναφέρεται θα έχουμε εντυπωσιακή μείωση όχι μόνο των νέων γεωργών αλλά γενικότερα των γεωργών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ μιλούμε για 10,7 εκατομμύρια από τα 500 και βλέπουμε ότι η ανάλυση αυτή παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον όσον αφορά το αν πιάνουν ε, τόπο τα χρήματα της ε, κοινή αγροτικής πολιτικής για την πίτευξη αυτού του στόχου, δηλαδή το πώς ε, θα κινηθούν οι μέλουσες γενναίες όσον αφορά την Ήπεθρο και τη Γεωργία. Θα πρέπει επομένως όλα αυτά να τα δούμε στο ευρύτερο πλαίσιο του δημογραφικού προβλήματος στην ε, Ευρώπη. Τι λέει ο Πράσινη Θα έχουμε χάσει ως Ευρώπη μέχρι το 2035 35 έως 40 εκατομμύρια από τον συνολικό πληθυσμό. Άρα θα πρέπει να δούμε ε, στο σύνολο τι θα κάνουμε και επιμέρους βέβαια για την ε, γεωργική πολιτική και να δούμε τι θα γίνει με τους νέους γεωργούς ε, που ασκούν αυτή τη δραστηριότητα τόσο σημαντική, τόσο σημαντική για το ευρωπαϊκό μοντέλο. Οπότε εδώ υπάρχουν σοβαρές συνέπειες για την ατμόσφαιρα, για το έδαφος, την βιοπικιλότητα που όλα αυτά τα εξασφαλίζει η Γεωργία. Ο κ. Σαρπάμα μας είπε ότι θα πρέπει να δούμε το ευρύτερο τοπίο και να δούμε πώς ε, ο στόχος θα αναβαθμιστεί ούτω ώστε να ε, εκταμιώσουμε σημαντικά ποσά. Πάντως σύμφωνα με την ανάλυση μέχρι τώρα όλα αυτά τα χρήματα δεν έχουν ωφελήσει οπότε έχουμε από την ε, εισηγήτρια, μια παρουσίαση. Ε, συμφωνώ με το σημείο 4, όπως μας τα είπε, δηλαδή πώς θα, εξασφαλιστεί ότι η Επιτροπή και τα κρατή-μέλη θα βελτιώσουν το σύστημα της αξιολόγησης, του ελέγχου, της εποπτείας για το τι γίνεται με όλους αυτούς τους ε, πόρους που πάνε προς τους νέους γεωργούς. Όμως αυτό το οποίο δεν έχει καταστεί σαφές για μένα είναι τα σχετικά με τη σχέση κόστους αποτελέσματος. Ε, για να δούμε και να αναλύσουμε γιατί δεν αποδίδει το σύστημα όπως θα όφιλε να αποδώσει. μας πει η Ευρωπαϊκή Αγορή τι γίνεται στα πλαίσια της μεταρρύθμισης της ΚΑΠ να μας πει αν υπάρχουν κάποιοι μηχανισμοί ούτω ώστε να καλύψουμε τις ε, ανησυχίες, τις υποδείξεις ε, του ελληνικού συνεδρίου. Δούμε πώς θα βελτιωθούμε. νομίζω ότι έτσι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τη λέει η συνθήκη της Ρώμης για να, τι, τη λέει, λέει ότι θα πρέπει να υπάρχει επάρκεια κλπ. Έχουν αλλάξει από τότε βέβαια τα πράγματα. Αλλά ακόμη και έτσι καταρτίζουμε τον προπολογισμό και τις προάλλες είπαμε τον πρόεδρο του Ελληνικού Συνεδρίου ποιες θα είναι για το 2018 προτεραιότητες και έχουμε την ετησία έκθεση. Ε, δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι ε, ασήμαντα τα πόσα και είπε ο ε, ότι θέλουν να ε, κόψουν κάποια χρήματα, θα δώσουν σε άλλες ε, προτεραιότητες. Ε, εγώ νομίζω ότι είναι προτεραιότητα σημαντική και είναι πολιτική. Όμως θα πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη το ότι άλλαξαν οι παράμετροι. Άλλαξαν τα πράγματα. Είναι δύσκολη η παγκόσμια συγκυρία. Θα πρέπει να συγκεράσουμε τη βιώσιμη ανάπτυξη με τους στόχους ε, τον ε, σχετικά με τους γεωργούς και να δούμε πώς θα έχουμε δαπάνες αποτελεσματικές για την επιτύχηση των στόχων. Νομίζω ότι θα πρέπει να κρατήσουμε τους νέους στην ε, Ήπεθρο. Από ό,τι φαίνεται δεν το έχουμε καταφέρει. Οπότε αυτά εγώ θέλω να πω για αυτή την συζήτηση που είναι πολύ σημαντική. Είναι κάτι που αφορά ευρύτερα θέματα γιατί επίσης είναι σημαντικό θέμα το τι γίνεται με την Ήπεθρο. Είναι χρήσιμο να προβληματιστούμε για να δούμε πώς θα προχωρήσουμε προς την μεταρρύθμιση, να δούμε πώς θα βελτιώσουμε την κοινή πολιτική, πώς μπορούμε να σώσουμε τα πιο σημαντικά και ταυτόχρονα να έχουμε τα νέα κριτήρια, να έχουμε περισσότερη αποτελεσματικότητα και να μπορέσουμε να πετύχουμε τους στόχους που έχουμε και άλλους πιο φιλόδοξους μεγαλύτερου βεληνικούς. Είναι καυτό το θέμα. Είναι καυτή επικαιρότητα. Και πρέπει να υπάρχει στο θεματολογιό μας, Πρόεδρε. Από την Επιτροπή, η κυρία, α, η επικεφαλής της Διεύθυνσης για τις άμεσες πληρωμές. Έχει το λόγο. Κυρία Πρόεδρε, κυρία Καλμπάχ, κύριε Ζουδικόφσκι, μέλη της Επιτροπής, κυρίες και κύριοι. Καταρχάς, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την ευκαιρία να αλλάξουμε απόψεις για το σχέδιο του εγγράφου εργασία για την ειδική έκθεση για τους νεαρούς γεωργούς. Προφανώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμφωνεί ότι ένα αποτελεσματικό εργαλείο υποστήριξη ε, των ε, νεαρών γεωργών αποτελεί επιφυλακτική ανάγκη και αυτό αποτελεί και κρίσιμο τμήμα όλη μα τη πολιτική. Στην τελευταία μεταρρύθμιση τη ΚΑΠΑ δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή στο θέμα αυτό. Το πεδίο εφαρμογή των εργαλείων ε, ανάπτυξη τη υπαίθρου διευρύνθηκε και τα νέα αυτά εργαλεία στον πρώτο πυλώνα άμα χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά. Είναι πρόσφατο, το 2015 ξεκίνησε. Δεν είχαμε ακόμα πολύ χρόνο να εξετάσουμε τα αποτελέσματα, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά το θέμα της ανανέωσης των γενναίων, που προφανώς χρειάζεται μακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα για να φανεί. Στον τομέα της γεωργίας δε, η, η ανανέωση των γενναιών αποτελεί ένα πάρα πολύ περιπλοκό ζήτημα. Δεν μπορούμε να το κοιτάξουμε α, ε, πέρα από την οικονομική κατάσταση και τις διαστατικές ε, αλλαγές και προφανώς και από την εθνική και την τοπική νομοθεσία. Ένα σημαντικό στοιχείο είναι η πρόσβαση στις ε, εκτάσεις, στη γη και η απόφαση μεταβίβασης των εκτάσεων από τους ε, ηλικιωμένους ε, αγρότες. Όπως σας είπα λοιπόν αυτό το μέτρο εισήχθη στην τελευταία μεταρρύθμιση της ΚΑΠ Πρόκειται για ένα επιπλέον το για τους νερούς αγρότες που για πρώτη φορά αναλαμβάνουν τέτοιες επιχειρήσεις για το πρώτο έτος, από το πρώτο έτος και για πέντε έτη κατά το όριο. Ένα θέμα το οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επανελειμμένα έχει τονίσει είναι ότι θα πρέπει να κοιτάξουμε μόνο τι πληρωμέ προ του νερού αγρότε στον πρώτο πυλώνα. Γιατί δώσαμε, για παράδειγμα, πρόσβαση προτεραιότητα σε εκθέσει βασικών πληρωμών. Άρα το θέμα αυτό αποτελεί ένα top-up. Οι επιδοτήσεις λοιπόν που λαμβάνουν οι νεαροί θα πρέπει να εξεταστούν στο σύνολό τους, στον πρώτο πυλώνα, στο δεύτερο πυλώνα και προφανώς και από τις εθνικές πολιτικές. Στην ε, ανάπτυξη της υπαίθρου τώρα είδαμε ότι υπάρχουν ε, ιδιαίτερε προδιαγραφές για την καθήρση των νέων ε. Υπήρχε το θέμα της μεταφοράς ε, στις γνώσεις, ασυμβουλευτικές υπηρεσίες, υπηρεσίες, υπηρεσίες διαχείρισης αγροκτημάτων, συνεργασία και το καθεξής για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 υποστηρίζουμε, σκοπεύουν να υποστηρίξουμε 175.000 νεαρούς αγρότες. Όπως είπα στον πρώτο πυλώνα ασφαλώς, το αποτέλεσμα των πολιτικών αυτών σε ό,τι αφορά την ανανέωση, την των γενναιών θα πρέπει να δοθεί συνολικά και μακροπρόθεσμα. Και για το μέλλον θα γίνει ενδελεχής ε, ανάλυση του αντικτύπου για την ανανέωση των γενεών. Θα γίνει αξιολόγηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία θα ξεκινήσει στα τέλη του 2017. Επίσης, όπως γνωρίζετε, στις 29 Νοεμβρίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα δημοσιεύσει την ανακοίνωση για το μέλλον των τροφίμων και της γεωργίας. Αυτή η ανακοίνωση θα δώσει ιδιαίτερη σημασία στην ανανέωση των γενεών και στην ανάγκη να υπάρχουν στόχοθετημένες δράσεις προς την κατεύθυνση αυτή. Και όπως είπατε, ο ρόλος των κρατών μελών και η διάδραση μεταξύ των διαφορετικών εργαλείων στον πρώτο και δεύτερο πυλώνα και η επικέντρωση στην απόδοση θα καλυφθούν επίσης από την ανακοίνωση αυτή. Αναφέρθηκαν και διάφορα συγκεκριμένα ερωτήματα από πλευρά των βουλευτών Καταρχάς, ε, ότι είναι αδύναμη η αξιολόγηση των αναγκών σε ό,τι αφορά το πρώτο πυλώνα. Όπως θα ξέρετε, η υποστήριξη εισοδήματος αποτελεί ένα γενικό μέτρο στήριξης. Θα πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη σημασία στην απλούστευση και θα πρέπει όλο αυτό να ακολουθήσει τη λογική των πληρωμών ε, πρώτο πυλώνα. Γενικές και απλές πληρωμές. Υπάρχει μεγάλος αριθμός δικαιούχων, 7 εκατομμύρια γεωργοί. Και η προσέγγιση μας δεν ήταν ποτέ να κάτσουμε να ελέγξουμε τον κάθε ετούντα για τις μεμονωμένες ανάγκες του, αλλά να παρέχουμε πιο πολύ γενική υποστήριξη στον τομέα αυτό, όπου φυσικά θα πρέπει το εισόδημα να συνάδει με την υπόλοιπη οικονομία. Επίσης, εισάγαμε ένα σύστημα όπου θα υπάρξει επιλογή έργων στον το σύστημα του πρώτου πυλώνα. Αλλά όλα αυτά προφανώς θα τα εξετάσουμε και για το μέλλον. Για το δεύτερο πυλώνα τώρα. Εδώ υπογραμμίζουμε το μεγάλο ρόλο που έχουν να παίξουν τα κράτη-μέλη στον προγραμματισμό τους, στο σχεδιασμό τους. Θα πρέπει να γίνει αυτή η ανάλυση σε πρώτη φάση για να ληφθούν υπόψη όλες οι καταστάσεις, όλα τα εργαλεία τα οποία εφίστανται σε τοπικό επίπεδο σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη της υπαίθρου, ο στόχος για την υποστήριξη των νεαρών αγροτών γίνεται μέσω κριτηρίων επιλογής. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δίνει αρρωγή προς τα κράτη-μέλη, συμβουλές, ε, αλλά προφανώς η αξιολογική των αναγκών θα πρέπει να γίνει από τα κράτη-μέλη. Ετέθησε και το θέμα του Omnibus ίσως να μην είναι το σωστό σημείο να σχολιάσουμε το Omnibus, αλλά μιας και το έθεσε ο κύριος Φλάνναγκαν, να σας πω ότι πλέον αυτή η υποστήριξη διτίθεται για περίοδο 5 ετών για όλους τους γεωργούς. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Δεν κατάλαβα ποιο είναι το σχέδιο της Κομισιόν ε, για την αλλαγή. Δεν κατάλαβα τι κάνουμε τώρα γιατί πραγματικά το ελεγκτικό συνέδριο ε, είναι πολύ συγκεκριμένο και πραγματικά ε, το να μας στέλνουν εδώ έναν επικεφαλής μονάδας, ο οποίος δεν μας λέει για την ε, πολιτική, τη γενική, δεν το καταλαβαίνω. Είτε θα έρθει εδώ λοιπόν ο Γενικός Διευθυντής, είτε ε, θα τα αφήσουμε όπως είναι. Αλλά γενικά δεν μπορούμε να εμφυσυχάσουμε. Δεν είναι προσωπικό, απλώς ε, δεν είναι δίκαιο. Για μια τέτοια ιστορία, για ένα τέτοιο θέμα, να παίρνουμε απαντήσεις σε αυτό το επίπεδο. Και υπάρχουν και άλλοι συνάδελφοι τώρα στο ημερήσια διάταξη, οι οποίοι θα ήθελαν να μιλήσουν με τον Γενικό Διευθυντή, κυρία Κάντενμπαχ. Ναι, συμφωνώ με την Πρόεδρο και την πρότασή της, γιατί έχω ε, για δύο πράγματα. Γενικά, ε, έχουμε εδώ σκοτάδι στην αίθουσα δεν βλέπουμε, βλέπουμε συνεχώς τις ίδιες απαντήσεις ε, για τα θέματα της γεωργικής πολιτικής. Είναι όλα η μαύρα ή η ασπρα Και δεν ξέρω ε, αν θα πρέπει να προσποιούμαστε απλώς ε, ότι δεν χρειάζεται να αλλάξει τίποτα ή να κάνουμε κάτι. Νομίζω ότι ο στόχος για το μέλλον της γεωργικής πολιτικής είναι και υψηλού επίπεδου τρόφιμα αλλά και υπηρεσίες και γεωργία βιώσιμη. Όλα αυτά πρέπει να τα διασφαλίσουμε, να διασφαλίσουμε τον ανταγωνισμό με άλλα προϊόντα και άλλες συνθήκες παραγωγής έτσι ώστε να χρησιμοποιούνται με τον καλύτερο τρόπο τα χρήματα των ε, φορολογουμένων. Δυστυχώς σε αυτή την έκθεση δεν έχω αυτή την εντύπωση. Την Δευτέρα έχουμε τον Επίτροπο Χογκάν με τον οποίο θα συζητήσουμε. Σας ευχαριστούμε λοιπόν για τις ε, ε, πληροφορίες. Ο κύριος Βατερχόφσκι στο τέλος έχει το λόγο. Ευχαριστώ τα μέλη του Κοινοβουλίου, τους ε, βουλευτές, τους κυρίους ε, Φλάναγκαλ, Σεβκέμψκη, Σαλαφράγκα, Σμιτ και τον την εκπρόσωπο της Επιτροπής. Εν συντομία, ένα ήταν το ερώτημα στη συζήτηση, το πρόβλημα της αξιολόγησης. Σήμερα το απόγευμα θα παρουσιάσω την επόμενη έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου για το πρόγραμμα, το προγραμματισμό της ε, αγροτικής ανάπτυξης και του προγράμματος αυτού. 4L, ε, πολύ large, πολύ μεγάλο, πολύ μεγάλο ε, το χρονικό διάστημα, πολύ αργά. Όλα αυτά τα στοιχεία τώρα που ξεκινάμε τη συζήτηση για το μέλλον της ε, γεωργικής πολιτικής είναι σημαντικά γιατί δεν έχουμε αξιολόγηση της προηγούμενης περίοδου. Σήμερα το απόγευμα θα δείξω ότι το 2017 μόνο 10% των προγραμμάτων για την γεωργική ανάπτυξη, την αγροτική ανάπτυξη δαπανήθηκαν. Πέρυσι ήταν 70%, φέτος μόλις 10%. Ξεκινάμε το σχεδιασμό του μέλλοντος, αλλά δεν έχουμε αξιολόγηση της προηγούμενης εφαρμογής. Η κυρία Κάντεμπαχ τώρα μίλησε για τους φραγμούς. Η βασική φραγμή, τα βασικά προβλήματα είναι η πρόσβαση στη γη. Οι περισσότεροι νέοι γεωργοί αυτό θέτουν ως πρόβλημα, την πρόσβαση στη γη. Το τελευταίο ερώτημα έχει το τελευταίο ζήτημα έχει ως εξή. Μην ερμηνεύσετε την έκθεσή μας ως πρόταση για μείωση των επιδοτήσεων των νέων γεωργών. Ποτέ να μην γίνει αυτό. Είμαι ο πρώτος που λέω ότι η Ευρωπαϊκή Γεωργία χρειάζεται υποστήριξη, αλλά πρέπει η στόχευση να είναι καλύτερη για να έχουμε πραγματικά αποτελέσματα. Το πρόβλημα των νέων γεωργών είναι πρόβλημα όχι μόνο οικονομικής υποστήριξης. Έχετε δίκιο, υπάρχουν και πολλές άλλες παράμετροι και πολλές άλλες λύσεις που μπορούν να δοθούν για να πετύχουμε αυτή την ανανέωση των γενεών. Είναι περίπλοκο το ζήτημα της ε, ε, οικονομικής υποστήριξης. Α, ε, και άλλη μία πρόταση και τελειώνω. Κυρίες και κύριοι, χρειαζόμαστε στη Γεωργία μια, ένα όρο, όραμα μια ενα οραμα μακρύ μακρυπνο μακρόπνο, όχι τρία-τέσσερα χρόνια. Γιατί η μείωση των κονδυλίων στα επόμενα 3-4 χρόνια, σε πόσες επιχειρήσεις, σε πόσες εκμεταλλεύσεις θα οδηγήσει τα επόμενα χρόνια, μικρές, μεγάλες εκμεταλλεύσεις, αυτό είναι πολιτική επιλογή. Ο σχεδιασμός του μέλλοντος της κοινή αγροτικής πολιτικής πρέπει να είναι μακρόπνος, όχι μόνο 3, 4, 5 χρόνια. Ευχαριστώ πολύ για τη δυνατότητα που μου δώσατε να παρουσιάσω αυτή την έκθεση. Η συνάδελφος Αγιάλα. Sí, solamente, es que justamente en relación a esto que acaba de decir... Ακριβώς είναι τα πράγματα όπως τα είπατε κύριε Βοητσόσκη. αυτό ήθελα και εγώ να πω ότι η μελέτη του Ελληνικού συνεδρίου ήταν ενδελεχής. Όπως είπατε, ξέρετε δεν είναι καν θέμα ότι κάνει άλλα, άλλα πράγματα σε κάθε, σε κάθε περιφέρεια διαφορετικά. Αυτό και στην Ισπανία. Υπάρχουν ε, ε, ιστορικοί λόγοι και ε, όλα εξαρτώνται τελικά από κάποιες νομοθετικές ε, ρυθμίσεις. Ε, είδατε γιατί έγινε στην Ελλάδα με το σύστημα της ε, μεταβίβασης κυριότητας. Οπότε θα πρέπει να δούμε το θέμα ανά περιφέρεια. No, this, this, question... Το ελληνικό συνέδριο. Ναι, αλλά αυτό δεν ήταν αντικείμενο του οικονομικού ελέγχου, γιατί η εθνική νομοθεσία δεν επιδέχεται οικονομικό έλεγχο. Συμφωνώ μαζί σας όμως ότι αυτού του είδους η προσβασιμότητα στην γη είναι σημαντική. Να, εκτός του ελέγχου τώρα να σας πω όφερα στην Πολωνία τελευταία φορά που είχαμε τροποποιήσει τις νομοθεσίες μπήκε όριο για το πόσο γη μπορεί να αποκτήσει κάποιος εάν δεν είναι υγιοργός. Άρα ευνοούνται οι γεωργοί. Να ένα παράδειγμα. Όμως αυτό δεν μπορούσαμε να το περάσουμε από τον οικονομικό έλεγχο, ήταν εκτός του αντικειμένου μας. Μάλιστα. Περιμένουμε και τη συζήτηση με τον Επιτροπό. Κυρία Κάτμπαχ, θέλετε το λόγο. Όχι. Ολοκληρώθηκε λοιπόν και το σημείο τη σημερινή διάταξη αυτό και το δημόσιο τμήμα της ακροασής μας. Θα σας παρακαλούσα να βγείτε από την αίθουσα ήσυχα και γρήγορα.